Meine... Αγαπητοί συνάδελφοι, παρακαλώ καθίστε. Κολλήγων, κολλήγων. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα να σας προσκαλέσω, να σας ε, χαιρετήσω, να σας καλωσορίσω καλύτερα στην συνεδρία στην απογευματινή μας. Πρέπει να συνεχίσουμε με το σημείο 15 που είναι το θέμα των σχέσεων με την Τινησία στο σημερινό περιφερειακό πλαίσιο. Και έχουμε την έκθεση του κυρίου Καστάλντο. Επιτρέψτε μου κύριε Καστάλντο να να καλωσορίσω το βραβείο τα βραβείο Σαχάροφ τα, τους βραβευμένους βραβείους Σαχάροφ που είναι εδώ και παρακολουθούν αυτήν την ε, συνεδρία και τον ε, εκπρόσωπο του κυρίου Αλ Μπαϊντάρη, ο οποίος είναι ακόμα στη φυλακή στην Σαουδική Αραβία. Να τονίσω ότι η κατάστασή του παραμένει η ίδια, ε, συνεχίζει να βρίσκεται στη φυλακή, αλλά θα δώσω στην κυρία Χάιντα το λόγο να, εξ ονόματός του να απευθυνθεί στην Επιτροπή μας. το λόγο.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 Σας ευχαριστώ για την παρουσία σας και για το κόπο που κάνετε να έρθετε εδώ. Ο κύριος Πονομάρεφ από τη Ρωσία επίσης. Θέλω και σας να σας ευχαριστήσω για τις προσπάθειές σας και τις προσπάθειες που κάνετε στην Ρωσία του ε, Πούτιν, ακόμα και στην εποχή του Μπρέσνιεφ ε, είχατε αγωνιστεί, επίσης το Σαλίτ Μαχμού, το Μοχαμετ που είναι από το Σουδάν που έχουν αγωνιστεί για την ε, ελευθερία της σκέψης και έχουν πάρει το βραβείο Σαχάροφ του 2007 η Σοφή Μπουσό επίσης που είναι εκπρόσωπος των δημοσιογράφων χωρίς σύνορα και θέλω και σας να σας ευχαριστήσω για το έργο του φορέα σας που είναι μεγάλη σημασία ακόμα και σήμερα στις ε, ημέρες αυτές στην Τουρκία την κυρία Άννα Λιβίνα που εκπροσωπεί την Λευκορωσική Ένωση των Δημοσιογράφων και ελπίζω ότι θα υπάρξει μια θετική εξέλιξη στη χώρα σας. Εν πάση περιπτώσει, προβλέπεται να γίνουν επαφές σε υψηλό επίπεδο. Η Τασλίμα Νασρίν η οποία ως δημοσιογράφος, ως συγγραφέας, ως ιατρός, ως ανθρωπίστρια έχει επιτύχει σημαντικά στον αγώνα κατά των διακρίσεων και των ανισοτήτων υποστηρίζοντας τα δικαιώματα των γυναικών και την ελευθερία της σκέψης. Χαίρομαι που είναι μαζί μας. Και χαιρόμαστε για το γεγονός ότι το βιβλίο που εκδώσατε είχε μεγάλη ε, κυκλοφορία και μεγάλη επίπτωση. Η κυρία Ζερεμπέγκοβιτς, ακτιβίστρια για τα ανθρώπινα δικαιώματα από το Σαράγεβο, η οποία από το 1998 έχει μεγάλη επιρροή με το έργο της ως δημοσιογράφος. Σας ευχαριστούμε λοιπόν που ήρθατε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και είναι μεγάλη χαρά που νιώθουμε που είσαστε μαζί μας. Λοιπόν, τώρα, τώρα μπορείτε να προχωρήσετε στα αραβικά. Έχετε το λόγο. مساء الخير أشكركم على إتاحتي هذه الفرصة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 لي Ήθελα να σας ευχαριστήσω. Είναι μεγάλη μου τιμή και μεγάλη ευτυχία που βρίσκομαι ε, εδώ μαζί σας και θέλω να σας μεταφέρω ένα μήνυμα από τον ε, σύζυγό μου, ο οποίος ε, βρίσκεται στη φυλακή εδώ και τρία χρόνια σας ε, μεταφέρω αυτό το μήνυμα και την έκκληση από τα παιδιά μου που έχουν στερηθεί τον πατέρα τους. Ένα μήνυμα ελπίδας θα να σας φέρω ώστε ο άνδρας μου μία μέρα να βρεθεί εδώ μπροστά σας, να έρθει να σας δει. Σας μεταφέρω επίσης και ένα μήνυμα ε, έκκλησης ε, για βοήθεια προς τον σύζυγό μου. Διότι η ελευθερία έκφρασης ε, είναι μια ελευθερία που πρέπει να απολαύουν όλοι οι άνθρωποι, άνδρες και γυναίκες, όλο τον κόσμο, ανεξαιρέτως. Επιτρέψτε μου πρώτα απ' όλα λοιπόν να απευθυνθώ εκ μέρους του συζύγου μου, του ΡΑΕΦ, από εδώ, από αυτή την ένδρα. Εγώ συχνά μιλάω για αυτόν και θα αξιοποιώ όλες τις ευκαιρίες, έχω αξιοποιήσει όλες τις ευκαιρίες που μου έχουν προσφερθεί το ίδιο πράττω και σήμερα. Θα ήθελα λοιπόν να του μιλήσω, να απευθυνθώ σε αυτόν κατευθείαν, να του πω όσα έχω στην καρδιά μου. Ραεφ, αγάπη μου, πριν από τέσσερα χρόνια βρέθηκαμε σε αυτό το άδειο διαμέρισμα. Άδειο διότι λείπεις. Και εγώ πρέπει να απαντώ τις ερωτήσεις των παιδιών, και εγώ διαρκώς ε, με, με απασχολεί το πώς θα συμπεριφερθώ όταν θα επιστρέψεις, θα κλάψω, τι θα σου πω. Τι θα κάνουμε, θα προετοιμάσουμε το βραδινό όπως συνήθως, ε, ε, θα κανονίσουμε τι θα φάμε, τι θα πιούμε, πώς θα αντιθούμε και συχνά αναρωτιέμαι ποιος είναι ο λόγος της μεγάλης οπουσίας. Είπα στα παιδιά που με ρωτούν συνέχεια ότι σου έχουν απαγορεύσει να ταξιδέψεις. Τα παιδιά μεγαλώνουν ε, συνεχώς με αυτό το ερώτημα και εγώ είμαι ευτυχισμένη διότι σου μοιάζουν. Έχουν το θάρρος σου, την ευφυΐα σου. Είσαι πιο ελεύθερος παρότι είσαι φυλακισμένος. Έχεις πολλούς φίλους ολόκληρο τον κόσμο πρέπει να σου πω. Ε, πολλές ε, ελεύθερες φωνές που μάχονται υπέρ της απελευθέρωσής σου. Οι συγγενείς σου, οι φίλοι σου, δεν είσαι μόνος σου. Δεν είμαστε μόνοι μας. Η αλληλεγγύη από πλευράς τους, η βοήθειά τους, η υποστήριξή τους είναι σημαντικές για μας. Θα ήθελα εκ μέρους σου να βοηθήσω για αυτή τη βοήθεια όλες τις ε, ελεύθερες φωνές στον κόσμο και ήθελα να πω εξ ονοματός σου Ραΐφ ευχαριστούμε όλους σας ευχαριστούμε και από πλευράς μου ευχαριστώ σας όλους Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ κυρία Χάιντα για τις πραγματικά πολύ εντυπωσιακέ κουβέντες σας ε, μια διακήρυξη αγάπης από πλευρά σας προς τον σύζυγό σας αλλά αυτό αποτελεί μια δήλωση και προς εμάς, ότι έχουμε το καθήκον να ε, αγωνιστούμε για τον άντρα σας και μάλιστα για όλους τους διακόμενους, για όλους όσοι ε, απέδειξαν το θάρρος και την τόλμη σας. Είπα στο συνεδριό σας ότι για μένα είναι αυτά εύκολα λόγια. Μπορώ να μιλώ όσο θέλω και σε καμία περίπτωση δεν θα φυλακιστώ και σε καμία περίπτωση δεν θα συμβεί κάτι κακό σε μένα για τα λόγια μου. το να είναι κανείς ε, Θαραλέο πολιτικός ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ε, προϋποθέτει πολύ θάρρος. Και αυτό νομίζω ότι είναι και η ουσιότητα διαφορά σας. Ευχαριστώ λοιπόν και εσάς και τον συνοδοιπόρο σας που είσαστε εδώ και να είστε βέβαιοι ότι θα είναι αυτό προτεραιότητα στη εργασία μας και κάποτε κάποιος είχε πει ότι ο άνθρωπος είναι ελεύθερος μόνο όταν είναι όλοι είναι ελεύθεροι. Σας ευχαριστώ πολύ λοιπόν που ήλθατε σε εμά σήμερα. So, wir fahren jetzt in unserer Tagesordnung. Και τώρα συνεχίζουμε στην ημερησία διαταξή, κυρίε και κύριοι. Με την έκθεση του εισηγητή μα, Καστάλτο, για την κατάσταση στην Τινησία στο παρόν ε, χρονικό πλαίσιο και έχουμε 27 τροπολογίες για την έκθεση. Ίσως να υπάρξουν και κάποιες συμβαστικές προτάσεις. Στις 13 και 14 Ιουνίου θα ψηφίσουμε στην Επιτροπή και το Σεπτέμβριο θα υποβληθεί στην Ολομέλεια η έκθεση, αν συμφωνείτε και εσείς ασφαλώς και έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα και εγώ να εκφράσω τις ευχαριστίες μου προς την κυρία Έντσα Φένταρ Μπαντάουι που μας έκανε την τιμή να βρεθεί εδώ σήμερα και να επαναπιβεβαιώσω την αμέριστη υποστήριξή μας για την απελευθέρωση του συζύγου τους στον οποίο έχει απονεμηθεί το βραβείο Σαχάροφ. Ε, το κοινοβούλιο μας πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες του και να τον ε, απελευθερώσει. Πρέπει να πάψει η δίωξη κατά των υποστηρικτών της Δημοκρατίας. Επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους που υπέβαλαν τροπολογίες ε, για την έκθεσή μου. Στη μεγάλη τους πλειοψηφία οι τροπολογίες αυτές είναι ιδιαίτερα επικοδομητικές αποδεικνύουν και το τεράστιο ενδιαφέρον που υπάρχει για την Τινησία αυτή τη στιγμή από πλευρά Επιτροπή ΑΦΕΤ. Να ευχαριστήσω και του σκιώδει συζητητέ με του οποίου μόλι τελείωσα μια πολύ επικοδομητική συνάντηση πριν από λίγο και οι οποίοι συμμετέχουν με μια προσέγγιση πολύ ανοιχτόμυαλη για την καλή πρόοδο των ε, διαπραγματεύσεων. Έχουμε υποβάλει 17 προτάσει συμβιβαστικέ που καλύπτουν τα κυριότερα σημεία τα οποία ε, εξετάζονται στην έκθεση γίνονται τεράστιες προσπάθειες σύγκληση από όλες τις πολιτικές ομάδες ώστε να καταλήξουμε σε μια έκθεση που να έχει την ευρύτερη δυνατή υποστήριξη. Είμαστε όλοι πεπισμένοι ότι την Ισία μπορεί και πρέπει να αποτελέσει μοντελό για τη Βορειοαφρική και για όλο τον Ισλαμικό κόσμο. Είναι κρίσιμη σημασία χώρα στην περιφέρεια αυτή και αποτελεί υπόδειγμα ε, διμερών σχέσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση. εγώ έχω ως σκοπό μια ευρεία συνένεση, ομόφωνη συνένεση μεταξύ των πολιτικών ομάδων που θα μπορούσε να αποτελέσει εφαλτήριο ε, διαπραγματευτικό όχι μόνο για μια εμπορική συμφωνία αλλά μια πραγματική συμφωνία πολιτικής εταιρικής σχέσης πολύ στενή ώστε η Τινησία να μετατραπεί στον μεγαλύτερο μας εταίρο με τη Βορεια ε, σύντομα έχουμε και άλλη ε, συνάντηση με τους κοιόδης συζητητές, οπότε δεν θέλω να σας κουράσω με άλλες τεχνικές ε, λεπτομέρειες που θα επιληθούν στη διάρκεια της συνάντησης αυτής με τους κοιόδης, αλλά θα ήθελα να εκμεταλλευτώ την ευκαιρία για να σας παρουσιάσω κάποια νέα στοιχεία ιδιαίτερα σημαντικά. Ειδικότερα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου προς το Κοινοβούλιο της ε, για τη νέα νομοθεσία περί κατανάλωση ναρκωτικών που πρότεινε η κυβέρνηση και που αυτή τη στιγμή ε, βρίσκεται υπό ανάλυση στην Ολομέλεια και που θα ρυθμίσει τις προβλεπόμενες ε, ποινές σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα για τα εγκλήματα αυτά. Έτσι όπως ζητήσαμε εμείς ε, ε, στη σχετική έκθεση και ε, όπως ε, επαναλαμβάνουμε στη συμβιβαστική πρόταση για μια πιο αποτελεσματική προσέγγιση στο θέμα της πρόληψης. Οπότε ελπίζουμε εκεί να επιτευχθεί ένα από το αποτέλεσμα σύντομα. Επίσης να αναφέρω συναδέλφους ένα σημαντικό πολιτικό γεγονός το περασμένο Σαββατοκύριακο έλαβε χώρα το 10ο συνεδρίο του ΝΑΤΑ όπου το 93,5 υπερψήφισε ένα ψήφισμα που διαχωρίζει την πολιτική από τη θρησκεία. Είναι πολύ σημαντικό ε, και θα ενισχύσει το ρόλο των ε, ε, κομμάτων τα οποία κόμματα θα μπορέσουν να συμβάλλουν στη δημοκρατική ζωή όλης της χώρας. κάτι που επιθυμούμε να συμβεί και στον υπόλοιπο Ισλαμικό κόσμο. Θέλαμε ειδικότερα να υπογραμμίσουμε και την ελευθερία του τύπου που ακούστηκε έντονα από διάφορους ε, συναδέλφους και αποτέλεσε αντικείμενο του συμβαστικής 3 και πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή επίσης και στους νέους όπως αναφέρεται στη συμβιβαστική 4. Επίσης, πολύ σημαντική ήταν κατά την απόψή μου η αναφορά στις πραγματικές και βαθιές αιτίες της ριζοσπαστικοποίησης ε, στη Συμβιβαστική 15, όπου αναφερόμαστε στον κοινωνικό αποκλεισμό, πράγμα το οποίο βέβαια θα αναλύσουμε και καλύτερα στην επόμενη συνάντηση που θα λάβει η χώρα την Πέμπτη μετά από την Ολομέλεια να ευχαριστήσω ξανά του συναδέλφου και ελπίζω ότι θα καταφέρουμε να ολοκληρώσουμε το συντομότερο δυνατό τη συζήτηση επί τη έκθεση. Θέλουμε να στείλουμε ένα χειρό μήνυμα υποστήριξη προ την Ισία. Ένα ε, μήνυμα πεποίθηση, απόλυτη πεποίθηση ότι θα στηρίξουμε τη δημοκρατική τη πρόοδο και, θέλουμε, και ότι θέλουμε να αποτελέσει εταίρο μα δημοκρατικό στην Ένωση ε, πραγματοποιώντα ένα πραγματικό ε, σημαντικό βήμα βάσει αυτή τη έκθεση κιόλα για να κερδίσουμε αυτή τη μάχη, την οποία στηρίζουμε τόσο πολύ εδώ στο Κοινοβούλιο. Ευχαριστούμε, θα μείνουμε στα Ιταλικά, διότι τώρα για το ΕΛΚ θα μιλήσει ο κ. Τσέζα και μετά ο κ. Παντζέρη για του ε, σοσιαλιστές. Δεν είναι τυχαίο που είμαστε όλοι Ιταλοί. Ήθελα να ευχαριστήσω τον κ. Καστάλντο για τι προσπάθειε που έχει καταβάλει για μια έκθεση η οποία είναι ιδιαίτερα ισορροπημένη και ειδικότερα για το πώς αξιοποίησε τη συμμετοχή όλων μας. Σήμερα έχουμε κάνει ένα επιπλέον βήμα σε σχέση με την περασμένη φορά που δοθήκαμε, συζητήσαμε, κάναμε μια γενική συζήτηση για την Τινησία και μετά μπήκαμε επί της ουσίας στις λεπτομέρειες. Ε, κάτι εξαιρετικό εδώ στο Κοινοβούλιο, ειδικότερα αν ε, σκεφτεί κανείς τι ακούσαν προηγουμένως ε, από την ε, σύζυγο εδώ που αναφέρθηκε σε αυτό το μήνυμα προς τον σύζυγό της. Είναι σημαντικό να κάνουμε τέτοια σημαντικά βήματα για να υποστηρίξουμε την ελευθερία και την υποστήριξη της δημοκρατίας. Αυτό χρειάζεται η Τινησία. Σε τέσσερι πυλώνε πολύ σημαντικού βασίζεται αυτή η έκθεση. Πρώτα απ' όλα στο γεγονό ότι πρέπει με πολύ συγκεκριμένο και αποτελεσματικό τρόπο να βοηθήσουμε την Τινησία για να προοδεύσει σε αυτή τη δημοκρατική διαδικασία η οποία οριμάζει αλλά συνεχίζει να χρήζει υποστήριξη με τρόπου όχι απαραίτητα μεγαλώσιμου. Χρειάζεται η Ευρώπη εδώ να κάνει μια συγκεκριμένη ε, δουλειά για να λειτουργήσει το κοινοβούλιο, οι κοινοβουλευτικέ ομάδε. Εγώ με συναδέλφου πήγαμε στην Τινησία και συναντηθήκαμε με του εκπροσώπου του κοινοβουλίου δεν ξέρουν πώς να λειτουργεί, πρέπει να λειτουργεί ένα κοινοβούλιο, πώς πρέπει να λειτουργούν οι ομάδες. Οπότε πρέπει να τους βοηθήσουμε να λειτουργούν πιο δημοκρατικά στο πλαίσιο των σημερινών κομμάτων στην Τινησία. Μετά υπάρχει ο άλλος πυλώνος, ο οικονομικός, ο οποίος συνοψίζεται στα εξής. Κάθε ευρώ που δαπανάτε, και σε αυτή την έκθεση περιλαμβάνονται πολλά στοιχεία για αυτό το θέμα. Κάθε ευρώ που δαπανάτε για την οικονομική ανάπτυξη της Τινησίας διασφαλίζει την ασφάλεια και στην Ευρώπη στο πλαίσιο, στο πολιτικό πλαίσιο βάσει των όσων πράγματα πάμε να κάνουμε στην Ισία. Υπάρχει το θέμα της ασφάλειας, το οποίο δεν μπορούμε να υποτιμάμε. Μην ξεχνάμε ότι σήμερα στην Τινησία υπάρχουν, ε, ζουν ένα εκατομμύριο Λίβοι, τους οποίους πρέπει να βοηθήσουμε όπως κάνουμε και στις άλλες περιοχές του κόσμου, στην Τουρκία και σε άλλες χώρες. Πρέπει να τις βοηθήσουμε, να τους βοηθήσουμε ώστε αυτά τα άτομα να ζουν με τρόπο αξιοπρεπή. Και πρέπει επίση να του βοηθήσουμε και σε θέματα ασφαλεία. Όλα αυτά περιλαμβάνονται στην έκθεση αυτή. Αναφέρομαι στη συγκινητικότητα, σε έρευνα, σε θεσμού, σε δομέ. Όλα τα ζητήματα αυτά είναι σημαντικά. Είναι αναγκαίο η πολιτική γειτονία να κάνει περισσότερα. Και σήμερα η Ευρώπη έχει πολλά εργαλεία τα οποία διαθέτει στις ε, χώρες της ε, για τους νέους και το ίδιο πρέπει να κάνει και για τους νέους της Τινησίας εργασία, σπουδέ, υποστήριξη του πολιτισμού στην Τινησία, διότι δυστυχώς ε, Δυστυχώ σήμερα σε πολλέ περιοχέ τη Τινησία υπάρχει μεγάλη ενεργεία και δυσαρέσκεια που πολλέ φορέ οδηγεί στην προσχώρηση τέτοιων ε, νέων ανθρώπων στην τρομοκρατία. Οπότε θέλω να ευχαριστήσω ξανά τον κύριο Καστάλντο για τι προσπάθειές του. Σήμερα κάναμε ένα βήμα προ τα εμπρό. Έχουμε 17 συμβιβαστικέ τροπολογίε. Τώρα υπάρχει κάποια ομοφωνία μεταξύ μα. αυτό είναι γεγονό. Ε, ήδη σε μερικέ εβδομάδε έχουμε κλείσει ε, τις δικές μας εργασίες και πιστεύω ότι με αυτέ τι εργασίε θα μπορέσουμε να συμβάλλουμε σημαντικά σε μια χώρα που πραγματικά καταβάλει τεράστιε προσπάθειε να ε, στηρίξει ζωντανή τη δημοκρατία. Ευχαριστώ. Αντώνιο. Κύριε Πρόεδρε, να υπογραμμίσω και εγώ το ότι οι προσπάθειες που καταβάλουμε είναι εξαιρετικές. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Ισηγητή για την πολύ σοβαρή του προσέγγιση και για τη διαθεσιμότητά του. Εγώ πιστεύω ότι η έκθεση αυτή αποδεικνύεται ότι θα γίνει πολύ σημαντική και ότι θα δώσει μια σαφή πολιτική γραμμή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Τινησία. Θα έλεγα ότι στόχος είναι να παρέχουμε όλα τα απαραίτητα εργαλεία τα οποία θα ευνοήσουν την ανάπτυξη της χώρας αυτής. Ειδικότερα δεδομένων των τρομοκρατικών επιθέσεων που έλαβαν χώρα και που αποτέλεσαν πρόσκομα για τον τουρισμό αλλά και για να φωθήσουμε με το θέμα της Λιβύης ε, που δυσχεραίνει τις ε, διάφορες δυνατότητες που υπάρχουν. Εμείς πρέπει να παίξουμε το δικό μας ρόλο και αυτό κάνουμε, επιλέγοντας την Τινησία ως πολιτική προτεραιότητα για να επενδύσουμε όχι μόνο πολιτικά αλλά και οικονομικά. Υπάρχει και μια έκκληση προς την Τινησία να παίξει και αυτή το δικό της ρόλο, προβαίνοντας σε μεταρρυθμίσεις και πιο συγκεκριμένα καθιστώντας ε, πιο ευέλικτη και ταχεία την νομοθετική δραστηριότητα, διότι πρόκειται για μια χώρα η οποία χρειάζεται άμεσα ε, οικονομικές και κοινωνικές μεταρρυθμίσεις. Τέλος, να υπογραμμίσω και εγώ το γεγονό ότι το πολιτικό πλαίσιο στην Τινησία, στην βρίσκεται σε ε, μεγάλη κινητικότητα και μια πτυχή σημαντική που ενδεχομένως δεν έχει ληφθεί επαρκώς υπόψη το συνέδριο του Ιαναντά που έλαβε χώρα πριν λίγες μέρες ε, μετα... είναι, ήταν επιλογή του Κανούση να διαχωρίσει την θρησκεία από την πολιτική δράση. Κάποιοι διεθνείς παρατηρητές λένε ναι μεν αλλά ε, είναι μια βιτρίνα μόνο από το κυβερνό κόμμα αλλά εγώ θα έλεγα το εξής ακόμη και αν πρόκειται για μια βιτρίνα δεν πάβει να ε, εδραιώνεται κατά κάποιο τρόπο η βούληση διαχωρισμού ε, μεταξύ πολιτικής βούλησης και θρησκείας και αυτό από μόνο του αποτελεί ιστορικό γεγονός το οποίο πρέπει να υπογραμμίσουμε και να ενθαρρύνουμε οπότε θα έλεγα από αυτή την άψη θα πρέπει να καταλάβουμε πόσο μεγάλη είναι αυτή η αλλαγή και να ενθαρρύνουμε την, την Ισία προς ε, την κατεύθυνση της μεγαλύτερης ανάπτυξης και της πολιτικής εξέλιξης. Πιστεύω λοιπόν τέλος ότι αυτή η έκθεση θα συμβάλλει πολύ σημαντικά. Ευχαριστούμε για τους συντηρητικούς ο κ. Μπασία. Πάρα πολύ σύντομα. Θέλω να ευχαριστήσω τους συναδέλφους μου για τις συναντήσεις των σκιωδών που είχαμε και ιδιαίτερα τον Φάμπιο, τον εισηγητή, για την προσέγγιση που είχε για τις διαπραγματεύσεις αυτές. Και πάλι η έκθεσή του σωστά διαρθρωμένη, με σωστή εστίαση και εύκολη, είναι εύκολα αναγνώσιμη. Βρισκόμαστε στο στάδιο των συμβιβασμών και υπάρχουν πολλές θέσεις που μπορεί να υποστηρίξει το κόμμα των συντηρητικών και μεταρρυθμιστών. Πρέπει να δώσουμε ένα μήνυμα υποστήριξης προς την Τινησία. Η οικονομική ανάπτυξη θα είναι και το υπόβαθρο της σταθερότητα και της ανάπτυξης <clears throat> και της ασφάλειας της Τινησίας. Οι θέσει απασχόληση για τον απλό πολίτη είναι το κλειδί. Και η παιδεία μπορεί να δημιουργήσει και τι ευκαιρίε για του νέου που θα του αποσπάσουν από τι ειρήνες του ριζοσπαστικισμού. Και μία σωστή μακροοικονομική αρρωγή μπορεί να βοηθήσει, αλλά θα πρέπει να συνδέεται με απτά ε, ωφέλη στο μικροοικονομικό επίπεδο. Δηλαδή μπορεί να φτιάξει κανεί αεροδρόμια, μπορεί να φτιάξει γέφυρες αλλά το να μπορέσει να αντιμετωπίσει την έλλειψη υδροδότησης και να δημιουργήσει γιατρούς και ε, εκπαιδευτικούς θα είναι πιο σημαντικό για τον απλό την Ισιο. Η κυρία... Ευχαριστώ. Θέλω να πω στον κύριο Καστάλτο, η κυρία το σχέδιο έκθεσής του είναι θαυμάσιο, είναι θαυμάσιο σε επίπεδο περιεχομένου και πράγματι εμφορείται από την φιλοσοφία που έχει διατυπώσει ο ίδιος. <clears throat> Θέλω να υπογραμμίσω αυτά που ελέγχθηκαν όλοι οι ομιλητέ μέχρι τώρα που εξηγούν γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να βοηθήσει την Ισία. Ένα θέμα το οποίο είναι ζωτικό και για την Ισία αλλά και για την Ευρώπη. Η Ισία είναι από τι λίγε, τι σπάνιε χώρε η οποία έχει ξεκινήσει και έχει προχωρήσει σε μια πραγματική δημοκρατική μετάβαση. Θυμόμαστε ότι και το βραβείο Νόμπελ της Ειρήνης έχει χαιρετήσει αυτήν την εξέλιξη. Ο κύριος Καστάλντι και ο κ. Πανσέλη τόνισαν την απόφαση του κόμματος Ενάντα για τον χωρισμό κράτους και εκκλησίας. Αυτή είναι μια απόφαση η οποία θα εισαχθεί και θα εδρεωθεί στα βασικά συνταγματικά κείμενα της Τινησίας όπου γνωρίζουμε όλοι πόσο μεγάλο πρόβλημα δημιουργούν η σύγχυση μεταξύ θρησκεία και κράτου σε πολλέ χώρε. Πρέπει να υποστηρίξουμε την θρησκεία στη δημοκρατική μετάβαση, να την υποστηρίξουμε γιατί διατρέχει μια οικονομική κρίση και είναι στα ύψη η ανεργία, ιδίω για του νέου και ιδίω στο νότιο τμήμα τη θρησκεία. Ξέρετε ότι ο τουρισμό είναι μια ένα από του αναπτυξιακού κλάδου στην Τινησία και δυστυχώ μετά τι τρομοκρατικέ επιθέσει έχει μειωθεί σημαντικά. Δεν είναι λοιπόν μοναχά θέμα ε, αλληλεγγύης. Είναι απαραίτητο να καταλάβουμε ότι είναι πολύ, πολύ σημαντικός ο τουρισμός για την οικονομική ανάπτυξη. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε και τα θέματα ασφαλείας, τις επιθέσεις, τον, <clears throat> τα σύνορα με τη Λιβύη, την αποσταθεροποίηση η οποία σοβεί στη Λιβύη αυτή τη στιγμή, το λαθρεμπόριο όπλων που κινείται και προς την Τινησία σε μεγάλο βαθμό, τον τεράστιο αριθμό προσφύγων που φεύγουν από τη Λιβύη και πηγαίνουν στην Τινησία με όλα τα συμπαρομαρτούντα για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η Τινησία. Πρέπει λοιπόν να βοηθήσουμε αυτή τη χώρα. Εγώ πιστεύω ότι η Ευρώπη έχει κάνει μέχρι στιγμής πάρα πολλά πράγματα. Το πρώτο τρίμηνο του 2016 έχουμε <clears throat> ψηφίσει πολύ σημαντικά κείμενα ψηφίσαμε το ψήφισμα για μια οικονομική και πολιτική εταιρική σχέση με την, ε, την και εγώ είμαι πρόεδρος της ομάδας παρακολούθησης για το θέμα αυτό που συνδυάσαμε πριν από λίγο. Ελπίζουμε ότι όλα αυτά πάνε προς, τα, προς την καλή κατεύθυνση. Επίσης έχουμε ψηφίσει μέτρα κατεπήγοντα για να υπάρξουν πρόσθετες ποσοστώσεις ελαιολάδου για την Τινησία και επίσης στην Επιτροπή Ίντα έχουμε εγκρίνει μια μακροοικονομική ε, βοήθεια 500 εκατομμυρίων ευρώ. Για το θέμα αυτό, το τελευταίο, όταν λέω ότι δόθηκαν αυτά τα πρόσθετα 500 εκατομμύρια, αυτά δεν είναι χορήγηση, είναι δάνεια που δίνουμε στην Τινησία. Η Τινησία όμως έχει ένα σημαντικό χρέος δεν είναι η πρώτη μακροοικονομική βοήθεια που τη δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση και επομένως θα πρέπει να δούμε κατά πόσο σε ευρωπαϊκό επίπεδο υπάρχουν κάποιες πρόπτικες όπως έκανε η Γαλλία και η Γερμανία να μετατρέψουν το, δα, το χρέος της ε, την Ισία σε αναπτυξιακά σχέδια τα οποία είναι πολύ σημαντικά για το μέλλον της χώρας και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να κάνει κάτι τέτοιο, γιατί αυτό είναι μια ρεαλιστική μορφή να βοηθήσουμε την ανάπτυξη στην Τινησία. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η κυρία Βερζιά έχει το λόγο τώρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε. Και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τον ε, συνάδελφο Καστάλτο για τον πολύ ευχάριστο τρόπο συνεργασίας και την αξιοποίηση των ευκαιριών για συμβιβασμού, για εξέβρεση συμβιβασμών που θα ικανοποιούν όλες τι πλευρές, γιατί είμαστε πεπισμένοι ότι όντω θα πρέπει να βοηθήσουμε την, την Ισία, γιατί είναι κρατικά σημαντική χώρα από πολιτικής άποψης, προκειμένου να υποστηριχθεί η δημοκρατική αυτή διαδικασία της ε, χώρας. Πολλά πράγματα έχουν προχωρήσει, ενδεχομένω όχι επαρκώ. Μία φίλη μου είχε εξηγήσει μετά την Αραβική Άνοιξη ότι και η Γαλλική Επανάσταση δεν ολοκληρώθηκε σε ένα χρόνο. Ενδεχομένω να, χρειαστούν λοιπόν ε, και πέντε χρόνια. Είναι μακρά δικασία, ξέρετε, η δημοκρατία και ο εκδημοκρατισμός. Αλλά φυσικά Υπάρχει και το κοινωνικό θέμα στην Τινησία, γιατί τα κοινωνικά ζητήματα δεν έχουν μετακινηθεί ούτε ρούπι από την ε, επανάσταση στην Τινησία. Η ανεργία, η φτώχεια, η Μαριέλτα ανάφερε όλα αυτά τα στοιχεία. Γενικά οι διαφορές, ε, οι οικονομικές, ε, ανεργία, σε ό,τι αφορά ιδιαίτερα το κομμάτι το νοτιοανατολικό της Τενησίας. Και για να απαντήσω σε αυτά που είπε η κυρία Δεσσαρνές, να πω ότι σε ό,τι αφορά την βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι σημαντικό η εταιρική σχέση αυτή να κινηθεί προς τη σωστή κατεύθυνση από οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο και η Ευρωπαϊκή Ένωση να μην προωθεί κάποια συγκεκριμένα συμφέροντα ε, εις βάρος των συμφέροντων της Τινησίας, γιατί θεωρώ ότι αυτό θα μας γυρίσει μπούμεραγκ σε τελική ανάλυση. Και ότι το θέμα αυτό στην παρούσα φάση προκαλεί ήδη σημαντική ζημιά στην Τινησία. Να τονίσω επίσης την ε, ανάγκη καταπολέμησης της τρομοκρατίας, γιατί την Τινησία αντιμετωπίζει σημαντικό πρόβλημα από αυτήν την άποψη. και στη χώρα αυτή. Όμως, ε, όπως και σε άλλες χώρες άλλωστε, δεν θα πρέπει να γίνεται αυτό ε, εις βάρος των βασικών θεμελιδών ελευθεριών που είναι ακόμα σε ευάλωτη θέση, όπως είναι η ελευθερία του τύπου, τα δικαιώματα των blogger κτλ. Και σε ό,τι αφορά το νομοσχέδιο κατά της δημοκρατίας, ε, ουσιαστικά διαπιστώνουμε ότι η Τινεσία ενίσχυσε την ποινή, τη θανατική. Δεν κινείται προς σωστή κατεύθυνση. Και το θέμα της μετανάστευσης είναι πάρα πολύ σημαντικό και θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι από τον πόλεμο στην ε, Λιβύη και μετά η Τινησία έχει υποδεχτεί ένα εκατομμύριο πρόσφυγες από τη Λιβύη και ούτε μόνο από τη Λιβύη, να το διευκρινίσουμε και αυτό, άτομα τα οποία διώκονταν στη Λιβύη. Ακριβώς το ίδιο δηλαδή, πως τη μία ποσότητα ανθρώπων, θέλετε, με αυτούς που κατέφθασαν ε, από τη Μεσόγειο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μιλάμε δηλαδή για ένα εκατομμύριο, έναντι δέκα εκατομμυρίων κατοίκους στην Τινησία, ενώ σε εμά ε, είναι ένα εκατομμύριο προς 500 εκατομμύρια, για να έχουμε έτσι μια αίσθηση μεγέθους. Και φυσικά αυτό έχει και οικονομικές ε, συνέπειες. Αυτό θα έπρεπε να σημαίνει και κάτι για την βοήθεια και τη χρηματοδότηση που δίνουμε στο Τενησιακό Κοινοβούλιο. Γιατί δεν διαθέτει του πόρου που χρειάζονται για να λειτουργήσει. Είναι πάρα πολύ σημαντικό επίση να υποστηριχθεί και η κοινωνία των πολιτών. Είναι σημαντικό να μην χρησιμοποιούνται οι πόροι τη Ευρωπαϊκή Ένωση προ την Τινησία για να αυξάνονται το χρέο τη Τινησία, το οποίο αυξήθηκε από 40 50%. τίφεται το θέμα της ε, ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών, τίφεται το θέμα της κινητικότητας. Ε. Και εμένα με ανησυχεί το γεγονός ότι βλέπω όλο και πιο πολλού νέους από το Μακρέπ και από την Τινησία να δυσκολεύονται να πάρουν βίζα για να έρθουν να σπουδάσουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρόκειται για συγκεκριμένα σημάδια και συγκεκριμένα σήματα, αν θέλετε, τα οποία αποστέλει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Χρειάζονται λοιπόν εξέλιξεις οικονομικές και κοινωνικές, αλλά δεν θα πρέπει να γίνονται εις βάρος της κοινωνίας και της οικονομίας και του πολιτισμού της Τινησία. Δεν θα πρέπει να γίνονται εις βάρος των επιχειρήσεων στην Τινησία και θα πρέπει να υποστηρίξουμε κάποια έργα ιδιαίτερα της κοινωνικής οικονομίας που ανθίστην την Ισία. Όλα αυτά λοιπόν μου φαίνονται πάρα πολύ σημαντικά. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, λέει ο πρώτα απ' όλα θέλω να χαιρετήσω το έργο, να εξάρω το έργο που έχει κάνει και ο συνάδελφός μας, ο κύριος Καστάλτος εισηγητής, αλλά και το σύνολο των συγγειωδών εισηγητών και συντακτών αυτής της έκθεσης. Νομίζω ότι έχουμε καταλήξει σε μια έκθεση η οποία επιτρέπει να καταδείξουμε το δρόμο που θέλει να ακολουθήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση προς την κατεύθυνση μιας ενίσχυσης, όπως είπανε πολλοί <clears throat> προλαλήσαντες, ενίσχυσης της βοήθειας που παρέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση στην Τινησία. Εγώ έχω μεταβεί στις 18 και 19 Απριλίου στο ΣΟΥΣ με μια πρόσκληση ε, φορέων τοπικών εκεί με την αιγίδα, υπό την αιγίδα του Πρωθυπουργού της Τινησίας και ήμασταν παρόντες σε μια συνέλεξη της ε, συνδιάσκεψης στο ίδιο ξενοδοχείο όπου τον Ιούνιο, τον προηγούμενο Ιόνιο υπήρξαν 38 θύματα των τρομοκρατών. Για μας λοιπόν αυτό σημαίνει ότι έχει ένα συμβολικό χαρακτήρα η παρουσία μας, γιατί καταδεικνύουμε με τον τρόπο αυτό ότι την Ισία είναι πάντα έτοιμη να αντιμετωπίσει αυτή την τρομοκρατική απειλή. Μετά από τις δύο αυτές ημέρες συνδιάσκεψης στο ΣΟΥΣ, είναι φανερό ότι η οικονομική κατάσταση είναι τρομερή. 80% των ξενοδοχείων στο μοναστήρ έχουν κλείσει ουσιαστικά από τον προηγούμενο Ιούνιο δεν έχετε πια κανένας Ευρωπαίος τουρίστας στην Τινησία. Είναι λοιπόν και αυτό ένα θέμα ανάκτησης της εμπιστοσύνης των Ευρωπαίων στην Τινησία και αυτό απαιτεί κάποια μέτρα ασφάλειας τα οποία έχουν να κάνουν με τα 500 και χιλιόμετρα συνόρων μεταξύ της Λιβύης και της Τινησίας. Ξέρουμε πόσο ασταθής είναι ακόμα η κατάσταση στη Λιβύη και εξακολουθεί να επηρεάζει αυτή η αστάθεια και την Τινησία. Γίνονται τρομοκρατικές επιδρομές στο νότιο τμήμα <clears throat> της ε, Τινησίας, κάτι το οποίο εκτρέφει μια πάρα πολύ σημαντική αβεβαιότητα και ανασφάλεια σε όλο το κράτος της Τινησίας. Επομένως, πέραν της οικονομικής βοήθειας που θα πρέπει εμεί να ενισχύσουμε από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα σε επίπεδο ασφαλείας, ώστε να ενισχυθεί ακόμα περισσότερο η ασφάλεια σε αυτό το κοινό σύνορο με τη Λιβύη και επίσης θα πρέπει να συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για να εξασφαλίσουμε την ενότητα του κράτους της Λιβύης γιατί μόνο σε αυτή την περίπτωση θα μπορέσει να εξασφαλιστεί και η ασφάλεια στις όμορες χώρες, μεταξύ των οποίων και την Ισία. Ευχαριστώ κύριο Γκάλερ. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Και εγώ τακτικά μεταβαίνω στην Τινησία από το 2013 και μετά και χαίρομαι λοιπόν που διαπιστώνω ότι υπάρχει ευρεία συνένεση εδώ στην αίθουσα. Να ευχαριστήσω και τον συνάδελφο Φάμπιο Καστάντο για το γεγονό ότι στην έκθεσή του ακριβώ αποτυπώνει αυτή την ευρεία συνένεση που επικρατεί στην Επιτροπή μα. Και πραγματικά αναφέρει όλα τα σχετικά στοιχεία στην έκθεση. Να τονίσω δε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι θα πρέπει να συνεχίσουμε να υποστηρίσουμε τους συναδέλφους μας, τους ομολόγους μας στο κοινοβούλιο εκεί. Γιατί πραγματικά έχουν μεγάλο καθηκόντων, το οποίο όμως θα πρέπει να είναι σε θέση να μπορούν να το ε, επιτελούν. Και χρειάζονται λοιπόν πόρους, χρειάζονται όλα τα απαραίτητα για να μπορούν να εκτελούν τα καθήκοντά τους αυτά. Και θα ήθελα να τονίσω και κάτι θετικό εκ νέου. Από την αρχή μιλούσα για το Ισλαμικό, όχι το Ισλαμιστικό κόμμα και προσοχή στη διαφορά. Γιατί έχω πάντα την εντύπωση ότι μια μεγάλη πλειονότητα στο κόμμα αυτό υποστηρίζει την πίστη ως ένα σύστημα αξιών, όχι σαν ένα πολιτικό πρόγραμμα ε, δράσης. Και νομίζω ότι στο συνέδριο που έγινε, συνειδητά έγινε αυτή η διάκριση. Και αυτό αποτελεί κάτι το φετικό το οποίο θα πρέπει να χαιρετήσουμε. Γιατί έχουμε πραγματικά συμφέρον το Ισλάμ να, συν, να συνάδει πολιτικά με τη δημοκρατία. Έχει πραγματικά συγκεκριμένα πρακτικά πλεονεκτήματα αυτό για μας. Και θα πρέπει πραγματικά να το αναφέρουμε ως κάτι θετικό. Προτάθηκε εδώ στην έκθεση, στον οικονομικό κλάδο, μεταξύ άλλων, να συμπεριληφθεί στο πρόγραμμα COSME η την Ισία για την αναγνωριστικότητα των επιχειρήσεων, το οποίο εστιάζεται ιδιαίτερα στι μικρομεσαίε επιχειρήσει. το καλωσορίζω αυτό ρητά. Επίσης, τονίζεται η ανάγκη μεταρρύθμισης του αγροτικού κλάδου. Αγαπητοί συνάδελφοι, όμως, θα πρέπει εφόσον και αν υποστηρίζουμε τη μεταρρύθμιση αυτή, στη συνέχεια να είμαστε και συνεπείς και ειλικρινείς και τίμοι, γιατί θα πρέπει στην περίπτωση αυτή να ανοίξουμε την αγορά μας για τα προϊόντα ε, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και αυτό θα πρέπει να αποτελεί κάτι αμφίδρομο. Δηλαδή η μεταρρύθμιση που θα γίνει, εάν ε, στεφθεί με επιτυχία, θα πρέπει να έχει και συνέπειες και θα πρέπει αυτό να έχει ενδεχομένω και αμοιβαία α, ωφέλη στο θέμα της ασφάλειας και της άμυνας τώρα. Θα πρέπει να κάνουμε μια σωστή ανάλυση μετά από διάλογο με τους ταινίσεους για το τι χρειάζονται και θα πρέπει να τους δώσουμε α, αυτά που χρειάζονται. Γιατί σε τελική ανάλυση είναι προπύργιο και δικό μας. Αν τα πράγματα πάνε στραβά εκεί, θα έχει επιρροή αυτό και σε εμάς. Τα δικά μας λοιπόν συμφέροντα θα προσπιστούμε με τον τρόπο αυτό και μην σας πω ότι είναι και πιο ευνοϊκό από οικονομικής άποψης αν φροντίσουμε ή την ίση να πετύχουν στον αγώνα τους κατά της τρομοκρατίας και κατά των υπόλοιπων απειλών. Και ως εκ τούτου υποστηρίζω λοιπόν και αυτές τις ε, πτυχές οι οποίες αναφέρονται στην έκθεση επί του συνόλου Είμαι πεπισμένος ότι θα είναι πολύ γύρω και θετικό το μήνυμα προς τους φίλους μας στην Τινησία. Θα τους δώσουμε μια ενθάρρυνση για τη τελική ανάλυση. Το κρατός θα πρέπει να είναι σε μια θέση, σε μια κατάσταση όπου ο κόσμος θα βλέπει ένα βίωνο μέλλον. Μια προπτική ανάπτυξη σε ένα καλοβιωτικό επίπεδο στην πατρίδα του. Σας ευχαριστώ. σα ευχαριστώ και πάλι ο κ. Καστάλτο τώρα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Είδατε, για σας. Για σας και μόνο. Έπρεπε να σας ζητήσει να απαντήσετε στα ρουμάνικα. Όχι, όχι, θα συνεχίσω στα ιταλικά, λέει ο κ. Καστάλντο. Όπως ακούσαμε και από τους διαφορούς συναδέλφους, έχει διαμορφωθεί μια κατάσταση που δεν είναι βέβαια κανόνας, αλλά θα μπορούσε να γίνει στο μέλλον. Ε, διαμορφώθηκε λοιπόν μια σύγκληση λόγω των διαφορών ευαισθησιών που έχουμε από κοινού και που καταφέραμε να συμπεριλάβουμε με τις προσπάθειές μας σε αυτή την έκθεση. Αντιλαμβάνομαι από όλες τις παρατηρήσεις που ακούσα από τους συναδέλφους ε, ειδικότερα όσον αφορά και την επανεκκίνηση της ανάπτυξης του τουριστικού τομέα που επλήγει σημαντικά από τις βίες επιθέσεις ε, των τελευταίων ετών. Θέλουμε λοιπόν να επανεκκινήσουμε και την εικόνα, να ανενώσουμε την εικόνα της Τινησίας, ε, την ε, αξιοπιστία, δεδομένων των τεράστιων προσπαθειών που έχει καταβάλει η χώρα στον τομέα τη ασφάλεια τα τελευταία χρόνια. Όλα αυτά είναι ύψη τη σημασία ώστε να καταπολεμηθεί η φτώχεια, η ανεργία, οι περιφερειακέ ανισότητε που αποτελούν ε, το θεμέλιο του κοινωνικού ζητήματο που αναφέρθηκε προηγουμένω. Είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα, ο μεγαλύτερο κίνδυνο ε, που αυτή τη στιγμή υπονομεύει τη δημοκρατική σταθερότητα τη χώρα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερος ε, και τους προλαλήσαντες, διότι κάναμε δουλειά που μπορεί να χρησιμοποιηθεί και εκτός του Κοινοβούλιου. Ε, ορισμένοι συμμετέχουμε στη μεικτή κοινοβουλευτική ε, Επιτροπή ε, για τις χώρες του Μαγκρέπ, την οποία προεδρεύει ο συνάδελφος κ. Παντσέρη και που μέσα στους επόμενους μήνες και τα επόμενα χρόνια θα ασχοληθεί με συγκεκριμένα ζητήματα, συγκεκριμένα θέματα που αφορούν συνεργασίες μεταξύ τη Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Τινησία και άλλων χωρών της Νότου τη Μεσογείου. Θεωρούμε λοιπόν ότι η δουλειά αυτή θα μπορέσει να δώσει μια οριζόντια ε, θεμελιώδη απάντηση κατά της ριζοσπαστικοποίησης και της τρομοκρατία, ώστε οι νέοι πράγματι να μπορούν να βρουν μια θέση απασχόλησης ε, σε τομείς ε, όπως αυτοί που αναφέρθηκαν όπως είπε ο συνάδελφος κ. Γκάλερ, στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, στο γεωργικό τομέα, στον τουριστικό τομέα που αναφέρθηκε ήδη, ε, τα ισχυρά ουσιαστικά σημεία της οικονομίας στην Τινησία. Ε, υπάρχει και ο συντονισμός με την Επιτροπή ΙΝΤΑ, με τις συνάδελφοντες Αρνές, ώστε να η έκθεσή μας να οδεύει παράλληλα με την πολιτική πτυχή ώστε να δώσουμε ένα ενιαίο ε, ηχηρό ε, μήνυμα στους συνομιλητές μας ε, σε όλους τους τομείς. Είμαι βέβαιος ότι θα συνεχίσουμε τη συνεργασία μας ότι αυτό να επιτευχθεί όπως πρέπει. Υποστηρίζω, όπως έγινε και στην Επιτροπή ΙΝΤΑ, υποστηρίζω λοιπόν στενάρα ότι είναι αναγκαίο ε, η μακροοικονομική υποστήριξη, η οποία μάλιστα εγκρίθηκε σήμερα με μεγάλη πλειοψηφία. Και φυσικά δεν αφαιρούμε την εστίαση για τα ζητήματα ασφαλείας. Θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντικό και το πρόβλημα της Λιβύης, όπου υπάρχουν σημαντικά προβλήματα ε, ε, για την επίλυσή του και μας ενισχύει ιδιαίτερα η δήλωση του στρατηγού Αφτάρ, ο οποίος για πολλωστή φορά απέρριψε την αναγνώριση της σημερινής ε, κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας, υπονομεύοντας το πολύ σημαντικό έργο του ΟΗΕ. Η σταθερότητα της Λιβύης σημαίνει σταθερότητα και στην Τινησία, σημαίνει σταθερότητα σε ολόκληρο το Μαγκρέμπ και σίγουρα αφορά και τη δική μας σταθερότητα, οπότε σε αυτό συμφωνώ απόλυτα με τα όσα είπε ο κ. Τσέζα Κάθε ευρώ που δαπανάμε για την οικονομική και κοινωνική πολιτική σταθερότητα της Τινησίας αποδίδει άμεσα ωφέλη και για εμάς. Αυτό ισχύει όχι μόνο για τις χώρες της Μεσογείου, όπου υπάρχουν πολλοί ε, Ιταλοί και Γάλλοι ε, συναδελφοί και αυτό μας ενδιαφέρει αλλά πρέπει όλα τα κράτη, ολόκληρη η να καταλάβουν ότι αυτό αποδίδει ωφέλη για όλη την Ευρώπη διότι έχουμε κοινά προβλήματα και κοινέ πρέπει να είναι και οι λύσεις. Ε, να εκμεταλλευτούμε λοιπόν αυτή την ιστορική ευκαιρία αφού αναφέραμε πολύ ε, αυτό το συνέδριο του Ισλαμικού Κόμματος ε, Χενάντα Α εκμεταλλευτούμε λοιπόν την ευκαιρία για να βρούμε και άλλου συνομιλητέ και να λάβουμε υποστήριξη από όλε τι ε, πολιτικέ ομάδε και στην Τινησία. Εμεί λοιπόν ω Ευρωκοινοβούλιο πρέπει να είμαστε οι πρώτοι που θα υποστηρίξουμε και τι κοινοβουλευτικέ εργασίε. Αληθεύει, όπω είπαν πολλοί, υπάρχουν πολλέ δυσκολίε στη λειτουργία των ομάδων. Ακόμη και σήμερα η χρήση ε, των οικονομικών μέσων που υπάρχουν ε, είναι ανεπαρκής για να χαρακτηριστεί δημοκρατικό και σύγχρονο κοινοβούλιο αυτό ενώ μιας δημοκρατικής και σύγχρονης ε, χώρας όπως η Τινησία. Θα πρέπει λοιπόν να δώσουμε κίνητρα και να ενισχύσουμε ακόμη και περισσότερο τις ε, δικές μας προσπάθειες προς αυτή την κατεύθυνση. Εκεί είναι πολύ σημαντικό και αυτό που γίνεται ε, στο ΔΕΚ και με ευχαριστώ και τον συνάδελφο κ. Γκάλερ που έχει αναλάβει ιδιαίτερε δεσμεύσει σε αυτό το μέτωπο με ένα ενιαίο μέτωπο θα, από εμά θα λάβουν την ίση ένα χειρό μήνυμα από εμά και με βέβαιο ότι συνεχίζοντα σε αυτή την οδό θα καταφέρουμε να του δώσουμε ακριβώ αυτό το μήνυμα. Ευχαριστώ και πάλι. Ευχαριστώ πολύ, λέει και ο πρόεδρο. Ούτω κλείνουμε τη συζήτηση για το θέμα τη θυνησία. Η ψηφοφορία θα γίνει τον Ιούνιο, 13, στις συνεδρίες 13 με 14 Ιουνίου και θα έρθει στην Ολομέλεια τον Σεπτέμβριο. Προχωρώ στο επόμενο σημείο της σημερινής διάταξης που είναι η παρουσίαση της μελέτης που ζήτησε η Επιτροπή μας στοιχεία για μια στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη σχέση με το Ιράν μετά από τη Συμφωνία για τα Πυρηνικά. Θα ήθελα να σας αναφέρω ότι η ύπατη εκπρόσωπος Μογκερίνη μετέβη στο Ιράν στις 16 Απριλίου μαζί με 7 επιτρόπους. Να σας πληροφορήσω ότι έχουμε και μια έκθεση ίδιας πρωτοβουλία για την, για την ε, στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς το Ιράν μετά την ποινική συμφωνία με τον κύριο Χάουτ ως εισηγητή και έχουμε ε, ζητήσει και μια μελέτη για τα θέματα αυτά για να προτείνει περαιτέρω ε, κατευθύνσεις για την σχέση Ευρωπαϊκής Ένωσης με το Ιράν. Οι συντάκτες της μελέτης είναι ο Δόκτωρ Ρουσμπεκ Παρσί, ο οποίος είναι ο Διευθυντής της ομάδα ερευνας Ευρώπη Ευρώπης-Ιράν στο Πανεπιστήμιο του Λούντ στη Σουηδία και την κυρία Διάννα Εσφαντιάρη που είναι ε, υπότροφη Μακάρθουρ στο King's College στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ο Δόκτωρ Πάρση είναι μαζί μας σήμερα και θα παρουσιάσει τα κύρια ευρήματα αυτή τη ε, μελέτη. Έχετε 10 λεπτά περίπου κύριε Πάση για να παρουσιάσετε αυτή τη μελέτη. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Να παρουσιάσω τα κυριότερα ε, πορίσματα αυτής της έκθεσης, αν θέλετε. Το κύριο στοιχείο αυτή τη έκθεσης, το κύριο στο οποίο καταλήγουμε, είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ιράν χρειάζονται να έχουν μια καλύτερη σχέση, μια πιο δομημένη σχέση μια πιο βιώσιμη μορφή διαλόγου μεταξύ τους και αυτό θα πρέπει να περιλαμβάνει και μια στρατηγική διάσταση. Όχι μόνο να είναι η επίλυση των των θεμάτων και των διαφωνιών, αλλά θα πρέπει να προχωρήσει περισσότερο για να έχουμε μια σχέση η οποία είναι πληρέστερη και επομένως <clears throat> πιο ανθεκτική και θα μπορέσει να ξεπεράσει τις αδίλητες και αναπόφευκτες πτυχές διαφωνιών το Ιράν έχει περάσει δύο σημαντικές εκλογικές διαδικασίες τα τελευταία χρόνια. Καταρχήν οι προεδρικές εκλογές που κέρδισε ο Ελ Ροχάνη τον Ιούλιο του 2013 και αυτό οδήγησε σε μια νέα πρωτοβουλία για την επίλυση του προβλήματος με τα πυρηνικά και αυτό ολοκληρώθηκε τον Ιούλιο του 2015 με την τελική συμφωνία. Επίσης φέτο τον Φεβρουάριο και τον Απρίλιο σε δεύτερο γύρο, έγιναν οι κοινοβουλευτικές εκλογές στο Ιράν, που ήταν σαφές ότι ο πληθυσμός εν γέννη και πάλι υπεστήριξε αυτούς που ήθελαν μια πιο ανοιχτή και καλύτερη σχέση με τη Δύση και με την Ευρώπη. Προς το παρόν λοιπόν μπορούμε να δούμε ότι υπάρχει η σωστή συγκυρία, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά το Ιράν, για μια καλύτερη και πιο βιώσιμη μορφή σχέσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η έκθεση συνεχίζει και αναλύει τις λεπτομέρειες και τις αρχές του διαλόγου που πρέπει να ακολουθήσει μεταξύ των δύο πλευρών. Το κλειδί εδώ είναι να διατηρήσουμε, τα, να λάβουμε υπόψη τα διδάγματα που, ε, που επέτρεψαν την επίλυση του θέματος αυτού του πυρηνικού, δηλαδή του κοινού σχεδίου δράσης, του JCPOA. Πρέπει να υπάρχει διάλογος ίσων και να υπάρξει συναντήληψη σε όλα αυτά τα θέματα. Αυτό είναι το βασικό πόρισμα. Δεν μπορεί να υπάρχει μια άνηση σχέση μεταξύ των δύο πλευρών. Η συνεργασία λοιπόν με το Ιράν είναι κάτι που να ξεπερνάει τη συνήθη διαδικασία των θεμάτων εμπορίου και επιχειρήν. Ασφάλεια ενεργειακή για την Ευρωπαϊκή Ένωση, προφανώς είναι σημαντική, αλλά και άλλα θέματα που η μεταλαμπάδευση τεχνολογία, οι ακαδημαϊκές ανταλλαγέ, η προστασία του περιβάλλοντος και η βιώσιμη ανάπτυξη. Όλα αυτά είναι το μισό και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει τεχνογνωσία και μεγάλο ενδιαφέρον και το Ιράν έχει την ανάγκη και γνωρίζει ότι η συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να είναι επωφελής. Υπάρχουν και τομείς τώρα διαφωνιών και μπορούν να υπάρχουν ε, επικρίσεις και από την Ευρωπαϊκή Ένωση προς το Ιράν και από το Ιράν προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά δεν είναι θέματα τα οποία πρέπει να λησμονηθούν ή να τα παραγνωρίσουμε, αλλά για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε, για να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε, να λύσουμε όλα αυτά τα θέματα ή για να καταλήξουμε τουλάχιστον σε μια κοινή κατανόηση ότι διαφωνούμε για τα θέματα αυτά, θα πρέπει να αντιμετωπιστούν τα ζητήματα αυτά μέσα σε ένα ευρύτερο πλαίσιο και μέσα σε ένα πλαίσιο το οποίο θα θεσπιστεί και πέραν του ύπατου πολιτικού επίπεδου. Για το λόγο αυτό θα προτείναμε να δημιουργηθούν ορισμένε ομάδε εργασία ή επιτροπέ εργασία με κρατικού αξιωματούχου και εμπειρογνώμονε και από τι δύο πλευρέ για να αντιμετωπίσουν αυτά τα συγκεκριμένα θέματα και όχι <clears throat> να γίνονται τα πάντα ένα θέμα πολιτική διαπραγμάτευση μόνο στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο. Υπάρχουν επίση τομεί κοινού ενδιαφέροντο, ιδίω σε ό,τι αφορά τα περιφερειακά ζητήματα, βλέπουμε την ανασφάλεια και αστάθεια στο Ιράκ και το Αφγανιστάν και φυσικά και το συνεχιζόμενο εμφύλιο της ε, Συρίας, όπου το Ιράν είναι ένας, από τους εμπλεκόμενους και όπου εν τέλει για να επιληθεί το πρόβλημα της Συρίας είναι απαραίτητο το Ιράν να συμμετάσχει στην Τράπεζα των Διαπραγματεύσεων. Όλα αυτά είναι τομεί όπου δεν συμφωνούμε κατά ανάγκη πάντα μας με το Ιράν. Αλλά εάν θέλουμε να επιληθούν όλα αυτά τα προβλήματα το Ιράν θα πρέπει να είναι παρόν στην τράπεζα των διαπραγματεύσεων και θα πρέπει να μιλάμε με το Ιράν και όχι απλώς να απευθυνόμαστε προς το Ιράν. Αυτά είναι λοιπόν μερικά από τα πιο σημαντικά θέματα όπου μπορεί να υπάρξει <clears throat> συνεργασία μεταξύ των δύο πλευρών και προσπάθεια επίλυσης θεμάτων και όχι μονάχα ε, αντιπαράθεση όπως το παρελθόν. Ένα περαιτέρω θετικό αποτέλεσμα από μια λύση των προβλημάτων αυτών θα είναι και η μείωση του αριθμού των μεταναστών και των προσφύγων που προσπαθούν να ξεφύγουν από τον πόλεμο και τη βία. Αυτό μας καταδεικνύει και πάλι ότι σε ό,τι συμβαίνει στην περιοχή αυτή, το Ιράν και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν κοινά συμφέροντα. Ό,τι συμβεί σε αυτή την περιοχή δεν επηρεάζει μόνο το Ιράν και δεν είναι μόνο το Ιράν ένα από του εμπλεκόμενου, αλλά είναι κάτι το οποίο θα επηρεάσει και την Ευρωπαϊκή Ένωση, επομένω είναι προ το στρατηγικό συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης να έχουμε ένα συνεχή διάλογο με όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές <clears throat> ώστε να μπορέσουμε να επηρεάσουμε την σύγκρουση αυτή που μας επηρεάζει με τη σειρά της όλους μας. Ευχαριστώ. Εμείς σας ευχαριστούμε. Ο κύριος Χαουίτ, ο εισηγητής, δεν είναι εδώ παρόν σήμερα. Οι συντονιστέ θα ήθελαν να πάρουν το λόγο. Ο κύριο Πρέντα. Θα θέλετε να πάρετε το λόγο και να πείτε δύο λόγια. Όχι. Ο κύριο Τάνοκ. Όχι. Άλλος κανείς. Ο κύριος Πιτέλα. Ο κύριος Μπούκνερ. Σας ευχαριστώ. Εγώ θεωρώ ότι υπάρχουν στην έκθεση αυτή κάποια προβλήματα. Στην σελίδα υπερθυμών 17, για παράδειγμα, αναφέρεται ότι το εμπόριο θα αυξήσει και θα βελτιώσει την ε, κατάσταση στην οποία διαβιώνει ο κόσμος στο, στη χώρα. Πιστεύω ότι το αντίθετο θα συμβεί, γιατί πρώτα θα πάρουν τα χρήματα αυτά Η πλήρη της Επανάστασης. Και λοιπόν, τα χρήματα αυτά θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν πιο πολύ για να καταπιεστεί προαιτέρω ο κόσμος. Πιο πολύ και από ό,τι σήμερα. Να προσέξουμε λοιπόν. Ίσως να είναι απεσιόδοξη αυτή η εκτίμηση, αλλά αυτό αποτελεί σίγουρα μία δυνατότητα, μία πιθανότητα την οποία θα πρέπει να λάβουμε υπόψη. Ας προσέξουμε λοιπόν στο σημείο 4 στη σελίδα 18 σε ό,τι αφορά τα περιβαλλοντικά ζητήματα. Εδώ αποτελεί μια μεγάλη καταστροφή και χρησιμοποιώ συνειδητά τον όρο καταστροφή του περιβάλλοντος της ε, λίμνης Ούνια. Είναι πραγματικά κάτι το οποίο αγνοεί παντελώς αυτή η έκθεση για την πυρηνική ασφάλεια. Υπάρχει ένας αντιδραστήρας ερευνητικό και υπάρχει συνεργασία μεταξύ των δυτικών κρατών και του Ιράν. Έχει ξεκινήσει αυτή η διαδικασία. Θεωρώ λοιπόν ότι χρειάζεται να γίνουν κάποιες διορθώσεις και κάποιες ευανθίτσεις σε κάποια από τα σημεία τα οποία πραγματεύεται η έκθεση. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Ο κ. Ποστινάρου έχει τώρα το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εγώ έχω μόνο δύο σύντομα σχόλια να κάνω, τα οποία αποτελούν και σημεία ανησυχία. Αφενό, θα πρέπει να προσέξουμε τον ρόλο που διαδραματίζει το Ιράν στην κρίση της Συρίας, ε, είτε είναι προ τα... προς το καλό είτε προς το κακό. Με το Ιράν θα πρέπει όλοι μας οι διάλογοι να εξερευνούν τις δυνατότητες να είμαστε ανοιχτοί με το Ιράν και να αναφέρουμε ότι οποιαδήποτε αρνητική επιρροή στην κατάσταση θα αποτελέσει λόγω ε, παγώματος των σχέσεων μας. Επίσης, υπάρχει ένα θέμα πιο ανησυχητικό σε ό,τι αφορά τα όπλα που είναι στα χέρια της Χεσμπολάχ. Και αν είναι επαρκή η συγκέντρωση των όπλων αυτών στα χέρια τη Χεσμολά και φτάνει σε ανησυχητικά επίπεδα, Ενδεχομένω να προκαλέσει ε, ρήξη μεταξύ διαφόρων ε, παραγόντων στην ε, περιοχή. Είναι ένα σημαντικό ζήτημα αυτό το οποίο θα πρέπει να το αντιληφθούμε και θα πρέπει να το συζητήσουμε ανοιχτά και με ειλικρίνεια με το Ιράν. Αλλά καλό είναι να μην ε, έχουμε ψευδεστήσει και αυτάπάτε στην παρούσα φάση. Θα είμαι αυτοκειμενική, Πραγματιστέ, αλλά θα πρέπει να θέσουμε επιτάπητο αυτά τα εξαιρετικά κρίσιμα ζητήματα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Μποστινάρου, άλλο κανεί. Από ό,τι φαίνεται δεν επιθυμεί να πάρει κανείς άλλο το λόγο. Έχετε το λόγο λοιπόν. Ευχαριστώ. Και θα ήθελα να απαντήσω στα θέματα αυτά για το εμπόριο με το Ιράν. Ότι αυτό βασικά θα ωφελήσει το RGC τους ε, ε, την επιστημονική φρουρά και όχι τον λαό του Ιράν. Αυτό είναι αρκετά απλοϊκό για το πώς λειτουργεί δηλαδή η οικονομία και η κοινωνία του Ιράν. Είναι σημαντικός πολιτικός παράγοντας αλλά η οικονομία του Ιράν είναι πολύ πιο πολύ σύνθετη. Δεν είναι στα χέρια μιας μικρής ομάδας ανθρώπων. Αυτό αφενός. Κατά δεύτερον, οι εμπειρίες μας από άλλε χώρες που έχουν υποστεί μαζικό εμπάργκο και κυρώσεις, είναι σαφές ότι ο μηχανισμός καταστολής του κράτους είναι ο τελευταίος ο οποίος επηρεάζεται από τις οικονομικές κυρώσεις. κοιτώντα το Ιράκ την δεκαετία του 90, ήταν σαφέ ότι όση πίεση και να ασκήσαμε στο Ιράκ, τότε ό,τι χρήματα είχαν ε, μείνει στα χέρια του Σαντάμ Χουσέιν πήγαιναν στο μηχανισμό καταστολής του κράτους. Καταλαβαίνετε λοιπόν σε ό,τι αφορά το RGC, ό,τι και να κάνουμε εμείς πάντα θα έχουν χρήματα στα χέρια τους. Το σκοπός του μεγαλύτερου εμπορίου με το Ιράν είναι ότι αυτό θα είναι υποφελές και για τη χώρα αλλά και για μας. Υποφελές για τη χώρα τι σημαίνει. Μικρότερη ενεργεία, πιο πολύ πλούτος για όλο τον κόσμο και πιο πολλοί τομεί αλληλεπίδραση μαζί μα. Αυτό δεν είναι τόσο, αν θέλετε, άμεσα πολιτικό ως ε, στόχος. Χρησιμοποιούμε την οικονομία για να έχουμε μεγαλύτερους τομεί αλληλεπίδρασης. Τώρα, το τι θα σημαίνει επακριβώς δεν ξέρουμε. Θα υπάρχει δηλαδή απαραίτητα μια μεταστροφή του κλίματος και μεγαλύτερη ευρωπαϊκή διάθεση. Όχι, δεν είναι σίγουρο αυτό. Αλλά το μόνο σίγουρο είναι ότι η απομόνωση ως τώρα ποτέ δεν έχει ωφελήσει τον οποιοδήποτε. Άρα ίσως θα έχει έρθει η στιγμή να δοκιμάσουμε μια διαφορετική οδό, μια διαφορετική μέθοδο για να υπάρχει διάδραση με πολλές άλλες ε, ομάδες και αυτό ελπίζουμε να έχει όφελος για την ε, κοινωνία, για την ε, Λίμνη Όρμια τώρα. Ναι, έχετε δίκιο, δεν την αναφέραμε γιατί θα μπορούσαμε να κάνουμε μια εξαίρεση, γιατί είναι μεγάλη η περιβαλλοντική καταστροφή που λαμβάνει η χώρα. Δεν είναι η μοναδική περιβαλλοντική καταστροφή, ξέρετε, απλά έχει λάβει τη μεγαλύτερη προβολή στον τύπο. Είναι πραγματικά μια ολόκληρη λίμνη που εξαφανίζεται, αλλά... Ε, αν θέλετε, από δυστατικής άποψης, η λίμνη αυτή είναι μόνο η κορυφή του παγόβουνου. Το βασικό πρόβλημα είναι ότι, για παράδειγμα, δεν υπάρχει ανακύκλωση ύδατο στη χώρα αυτή. Σε μια χώρα όπου η τροφοδοσία με νερό είναι πάρα πολύ ε, αβέβαιη και υπάρχει μαζική αστικοποίηση επί τρεις δεκαετίες χωρίς ε, την απαραίτητη πολεοδομία και χορταξία. Ε, απερίμωση επίσης στη χώρα. Υπάρχουν λοιπόν διαρθρωτικά δομικά ζητήματα τα οποία αποτελούν προβλήμα εδώ και πολύ καιρό. Τώρα όμως σιγά σιγά φτάνει κομπό στο χτένι και έτσι υπάρχει μεγάλη λειψιδρία σε πολλά μέρη και πολύ μεγάλη εξάρτηση από τις εποχιακές ε, βροχές, ε, βροχοπτώσεις, προκειμένου να βγάλουν τη χρονιά μέχρι τον επόμενο χειμώνα. Ναι, σημαντική λοιπόν και η λιμνιέρμια, αλλά υπάρχουν πολύ πιο πιεστικά, κατεπήγοντα περιβαλλοντικά προβλήματα. Η περιβαλλοντική τεχνολογία των ευρωπαϊκών χωρών που έχουν αναπτύξει ευρωπαϊκές χώρες θα μπορούσαν να ωφελήσουν εξαιρετικά τις πόλεις και την Ήπεθρο στο Ιράν. Τώρα, σε ό,τι αφορά το ρόλο του Ιράν στη Συρία, σε ό,τι αφορά τη Ναι, πιστεύω ότι το θέμα εδώ δεν είναι ότι προσπαθούμε να αποκρύψουμε τις σχέσεις ισχύω που υπάρχουν στην περιοχή. Σχέσεις ισχύω οι οποίες ε, κατά την άποψη πολλών κρατών μελών είναι επιβλαβείς για τη σταθερότητα στην περιοχή. Το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι να υπάρχει ένας στρατηγικός βιώσιμος, διαρκής διάλογος με το Ιράν να λάβουμε υπόψη τι θεωρούν αυτοί ότι αποτελεί εθνικό συμφέρον τους. Γιατί το να λάβουμε υπόψη το εθνικό συμφέρον τους δεν σημαίνει ότι αναγνωρίζουμε ότι έχουν δίκιο, ότι υποχωρούμε. Σημαίνει ότι υπάρχει μία λογική στον τρόπο άσκηση της πολιτικής τους. Και αυτό δεν έχει να κάνει με το να μας ενοχλούν εμάς, δεν θέλουν να μας την παίρνουν εμάς. Έχουν να έχει να κάνει με το πώς αντιλαμβάνονται τις απειλές, και τους κινδύνους για τη χώρα τους. Δεν σημαίνει ότι συμφωνούμε, αλλά ότι μπορούμε να τα λάβουμε αυτά υπόψη στις συζητήσεις μαζί τους. Γι' αυτό λοιπόν μιλάμε καταρχάς για ένα διάλογο μεταξύ ίσων, όχι για σχέσεις ε, πατεναλιστικές. Αν θέλουμε να τους πούμε τι πρέπει να αλλάξουν στη συμπεριφορά τους για να τους αναγνωρίσουμε, ε, ουσιαστικά αυτό θα αποτελέσει σίγουρα διέξοδο, γιατί δεν πρόκειται να συμβεί κάτι τέτοιο. Δεν θα κάτσουν να τους πούμε τι να κάνουν. Και αυτό είναι ένα από τα βασικά μαθήματα, διδάγματα που μπορούμε να αντλήσουμε από τις διαπραγματεύσεις για την επεξεργασία ενός κοινού προγραμματός εργασίας, όσο δεν λαμβάνουμε υπόψη τις προτεραιότητες τους, τις αντιλήψεις τους, δεν λέω να συμφωνούμε, αλλά να τις λαμβάνουμε υπόψη. Όσο θα το λαμβάνουμε υπόψη, δεν θα οδηγήσουν πουθενά οι διαπραγματεύσει. Το μοναδικό, ο μοναδικό κλάδο όπου πραγματικά υπήρχε αμοιβαιότητα, πραγματική όμω αλληλοαναγνώριση των αναγκών, ε, εκεί μόνο ευοδοθήκαν οι διαπραγματεύσει. Ευχαριστώ πολύ. Θα περάσουμε τώρα στο επόμενο σημείο στην ημέρα για διαταξή μας. Κοινή συζήτηση για την εταιρική σχέση και συμφωνία συνεργασίας Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκμενιστάν, σημεία 17-18. Η κυρία Ραμόνα Μονέσκου είναι η συγγήτριά μας. Αυτό είναι η συνέχιση της ε, συζήτησης που έχουμε κάνει στο παρελθόν για αυτή τη συμφωνία. Με 186 τροπολογίες που έχουν κατατεθεί, κάποιες από τις οποίες ζητούσαν να αναβληθεί η κύρωση της Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας. Η συγγήτρια, από ό,τι ξέρω, συμφώνησε με τους Χιώδης για ένα τρόπο να προχωρήσουμε που περιλαμβάνει μια νέα έκθεση η οποία θέτει ορισμένα ρεαλιστικά benchmarks που είναι απαραίτητο να επιτευχθούν προτού δώσει το Κοινοβούλιο την έγκρισή του. Χαιρετίζω την παρουσία του κύριου Τόιβο Κλάρ, που είναι ο επικεφαλή του Τμήματο Κεντρική Ασία τη Υπηρεσία Εξωτερική Δράση και θα λάβει το λόγο αργότερα. Αλλά προηγουμένω θα δώσω το λόγο στην κυρία Ραμόνα Μανέσκου για να παρουσιάσει την εκθεσή τη. Δεν ήσασταν η Ραμόνα Μανέσκου, από ό,τι καταλαβαίνω. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω τη γραμματεία της ΑΦΕΤ και τους σκιώδης συζητητές για την πολύ καλή συνεργασία που είχα μαζί της και τη βοήθεια που μου έχουν δώσει σε αυτό το έργο. Θέλω να ευχαριστήσω και τον εκπρόσωπο της Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης για την βοήθεια και τις πληροφορίες που μου έδωσε η υπηρεσία αυτή. Ήταν πάρα πολύ αποτελεσματική λοιπόν η συνεργασία μαζί τους. Θέλω επίσης να διαβεβαιώσω την Υπηρεσία Εξωτερική Δράση ότι τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, παρά το γεγονό ότι έχουν πάρει την απόφαση που έλαβαν ω σκιαγητέ, θέλουν να, συν, να συνεργαστούν μαζί σα και να συνεχίσουν τι βοήθειε, τι προσπάθειε για την βελτίωση του τη κατάσταση ανθρωπίνων δικαιωμάτων και κράτου δικαίου στο Τουρκμενιστάν. Ανεξάρτητα από την προσπάθεια που έχει γίνει ήδη από την Υπηρεσία Εξωτερική Δράση, σα υποστηρίζουμε. Όπως ξέρετε τώρα κύριε Πρόεδρε, λόγω των τροπολογιών που έχουν υποβληθεί και μετά από τη συζήτηση και την πρώτη ανταλλαγή απόψεων που είχαμε με, την, με τον κύριο Κούριαν, τον νέο ειδικό εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μετά από την συνάντηση που είχαμε ως σκιώδης συζητητές και εγώ, υπήρξε μια σαφής πλειοψηφία που ζήτησε να εγκριθεί η θετική γνωμοδότηση της ε, Επιτροπής μας για την Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας. Γι' αυτό ε, πήραμε μια πιστεύω σόφρονα απόφαση, ζήτησα από το Προεδρείο της ε, Επιτροπής μας να αναστείλει προσωρινά το περιεχόμενο αυτής της σύστασης μέχρι ότου διαμορφωθεί μια σαφής συνένεση <clears throat> στην Επιτροπή ΑΦΕΤ, ώστε να μπορέσουμε να εγκρίνουμε, να ψηφίσουμε θετικά για τη Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης και Σύνδεσης. Γιατί αυτό ήταν και το μήνυμα άλλων των πολιτικών ομάδων. Θέλουμε να ψηφίσουμε υπέρ, θέλουμε να δώσουμε την έγκρισή μας, αλλά κάτω από ορισμένε προϋποθέσεις που θα βοηθήσουν τις μεταρρυθμίσεις στο Τουρκμενιστάν. Συγχρόνως ζήτησα να ξεκινήσει και μια χωριστή διαδικασία που θα επιτρέψει στο Κοινοβούλιο να εκφέρει γνώμη σε σχέση με τη Συμφωνία Εταιρική Σχέση και Συνεργασία και θα είναι μια ενδιάμεση έκθεση η οποία βάσει του άρθρου 99,3 του κανονισμού του Κοινοβουλίου θα μπορέσει να έχει ένα περιεχόμενο που θα περιλαμβάνει βασικά στοιχεία τα οποία συμφωνήθηκαν μεταξύ των σχεδόν εισηγητών και μου της ίδιας όπως τα μέτρα που πρέπει να λάβουν οι αρχές του Τουρκμενιστάν σε σχέση με το κράτος δικαίου και τα ανθρώπινα δικαιώματα και να γίνουν μεταρρυθμίσεις στα θέματα αυτά. Ένα επίσης λειτουργικό μηχανισμό εποπτείας που να περιλαμβάνει συγκεκριμένα στοιχεία που θα πρέπει να δίδεται από την πλαίσια εξωτερική δράσης αναφορά για τα θέματα αυτά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και για να ξεκινήσουν οι διαδικασίε για να δημιουργηθεί μια πλήρη αντιπροσωπεία τη Ευρωπαϊκή Ένωση στην Ασκαμπάντ, κάτι που θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό και το οποίο θα δώσει και υποστήριξη για την επίτευξη του στόχου μα. Αν λοιπόν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εγκρίνει αυτό το ψήφισμα επί τη βάση μια ενδιάμεση έκθεση, θα μπορεί η Επιτροπή μα να ε, αναλύει περιοδικά την εκπλήρωση αυτών των κριτηρίων και να την αξιολογεί και αν η πρόοδος θεωρηθεί ότι είναι επαρκής, τότε η Επιτροπή μας μπορεί να επανακινήσει τη διαδικασία έγκρισης της Συμφωνίας Συνεργασίας και Εταιρικής Σχέσης με μια θετική ψήφο, κάτι που όλοι θεωρούμε ότι είναι ευκταίο και απαραίτητο. Περιμένουμε λοιπόν την απόφαση του διευρυμένου Προεδρείου της ΑΦΕΤ, που πιστεύω θα συνεδριάσει σήμερα Γνωρίζω ότι η Γραμματεία έχει διανύμει και μια επιστολή από τους σκιοδησιητές. Είμαστε όλοι καλώς πληροφορημένοι για τα θέματα αυτά. Τώρα για το περιεχόμενο αυτής της ενδιάμεσης έκθεσης εγώ θα συνεργαστώ με τους σκιοδησιητές και ο στόχος μας είναι να συμφωνήσουμε για το περιεχόμενο αυτής της έκθεσης. Θέλω να υπογραμμίσω επίσης την ε, προσπάθεια που έχει κάνει ο εκπρόσωπος της υπηρεσίας ε, εξωτερικής δράσης έναντι των αρχών της, του Τουρκμενιστάν, θα πρέπει να αναγνωρίσουμε τα θετικά βήματα και τα επιτεύγματα που έχουν λάβει χώρα μέχρι στιγμής. Ένα θετικό σημείο είναι και το γεγονός ότι το Τουρκμενιστάν έχει εγκρίνει το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα για το 2016-2020 με την υποστήριξη και τη βοήθεια εμπειρογνωμόνων των Ηνωμένων Εθνών. Αυτό μας καταδεικνύει <clears throat> ότι υπάρχει θέληση πολιτική και υπάρχει επομένω η ελπίδα να κάνουν περισσότερα, ακόμα περισσότερα οι αρχές του Τουρκμενιστάν. Γι' αυτό εγώ προσβλέπω στην ε, λήψη μιας απόφασης σήμερα από το διευρυμένο Προεδρείο της Επιτροπής μας και πιστεύω ότι πρέπει να συνεχιστεί συνεργασία και με τους και εισηγητές και με τον εκπρόσωπο της υπηρεσίας εξωτερικής δράσης ώστε να μπορέσουμε να προχωρήσουμε περισσότερο και να φτάσουμε κάποια στιγμή στην ε, φάση που θα μας επιτρέψει να εγκρίνουμε τη Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας με το Τουρκμενιστάν. Ευχαριστούμε. Τώρα, σύμφωνα με τους κανόνες μας, ε, σκιώδη συγγητέ είναι αυτοί που θα πρέπει να μιλήσουν. Μόνο ένα συναδελφό δικός μας είναι σκιώδη εισηγητής, ο κύριος Μπετίνη. Δεν ξέρω αν θέλει το λόγο. Ναι, παρακαλώ. Είστε ο μόνος που βρίσκεστε εδώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Σιγητρία, την κυρία Μανέσκου, διότι πραγματικά ε, είχε να ασχοληθεί με μια περίπλοκη πολιτική κατάσταση και επιτέλεσε ένα ε, εξαιρετικό έργο λαμβάνοντας υπόψη και τις ε, προτάσεις τροπολογιών συμβαστικών από τις διάφορες πλευρές και λαμβάνοντας υπόψη και τις διάφορες παρατηρήσεις που διατυπώθηκαν στη συζητήση μεταξύ των διαφορών ομάδων. Το ζήτημα είναι πολύ απλό. Όλοι θέλουμε να καταλήξουμε στην έγκριση αυτής της Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας. Ωστόσο, η έγκριση αυτή θα πρέπει να συνδεθεί με μια αποτελεσματική, ορατή βελτίωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε μια χώρα όπου το ζήτημα των ανθρώπινων δικαιωμάτων ακόμα εκρεμεί δραματικά. Όσον αφορά τις ελευθερίες τύπου, γνώμης της ε, ε, ελευθερίας των πολιτών ε, το Τουρκμενιστάν βρίσκεται στο τέλος των ταξινομήσεων παγκόσμια. Το κείμενο λοιπόν εμείς που προσπαθήσαμε να έχουμε, για το οποίο τελικά έχουμε καταφέρει να συμφωνήσουμε, αποτελεί μια λύση αρκετά απλή. θα πρέπει να ορίσουμε για το Τουρκμενιστάν ορισμένους στόχους επαληθεύσιμους, πολύ συγκεκριμένους, οι οποίοι θα μπορούσαν να μας δώσουν ένα σήμα ότι το Τουρκμενιστάν όχι έχει λύσει όλα τα προβλήματα, γιατί φυσικά αυτό είναι μη ρεαλιστικό, αλλά ότι τουλάχιστον ε, κάνει μια σοβαρή προσπάθεια σε πράξεις και όχι μόνο στα λόγια, μέσω, ούτε μέσω νόμων που δεν εφαρμόζονται ποτέ, Πρέπει λοιπόν να μπορούμε να επαληθεύσουμε με το τον τρόπο ότι το Τουρκμενιστάν έχει κάνει συγκεκριμένα ρεαλιστικά βήματα προς τα εμπρός. Δεν ζητάμε ε, πράγματα αδύνατα, απλά να βελτιωθεί η ζωή ανθρώπων που υποφέρουν, αρχές που ε, συμβολίζουν, θα συμβολήσουν την ε, ανανέωση αυτής της χώρας. Αυτή η πρόταση λοιπόν αναστολή δεν σημαίνει ότι τα τεινάζουμε όλα στον αέρα, αλλά ότι απλά θα παγιώσουμε μια ε, διαδρομή η οποία θα βοηθήσει την υλοποίηση των όσων ανέφερα. Συμφωνώ λοιπόν εγώ με τη θέση της συγκήτριας και εύχομαι μέσω της συνεργασίας με την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης να μπορέσουμε να παγιώσουμε αυτή τη διαδρομή στην οποία μάλιστα η υπηρεσία εξωτερική δράσης έχει ως καθήκον και θέτει ω στόχο να ε, κάνει συγκεκριμένα πράγματα όπως την αποστολή μιας αντιπροσωπείας στο Τουρκμενιστάν από την Ευρωπαϊκή Ένωση κάτι που έχει ήδη συζητηθεί και αυτό είναι ένας στόχος που έχουμε θέσει το χρονοδιάγραμμα είναι δύσκολο να το προβλέψει κανείς για τις εργασίες αυτές, αλλά θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε αμέσως, ώστε να έχουμε το συντομότερο δυνατό τα επιθυμητά αποτελέσματα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Μέζερης, παρακαλώ. Uh, Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πρόεδρε και ζητώ συγγνώμη προς, τον την εισηγητρία για το γεγονό ότι δεν ήμουν εδώ εξ αρχή. Ξέρω όμω ποια είναι η τοποθέτησή τη, γιατί το έχουμε συζητήσει επισταμένω στι διάφορε συναντήσει και προφανώ υποστηρίζουμε την εισηγήτρια για την απόφαση. Αυτό που θα πρέπει να διευκρινίσουμε, αλλά εξαρτάται πιο πολύ από το διαβριμένο Προεδρείο και όχι τόσο από την συνεμερινή συνεδρίαση, είναι το ποιο θα πρέπει να είναι το κείμενο για την ενδιάμεση έκθεση και κατά πόσο η έκθεση θα πρέπει να χρησιμεύσει ως βάση για τις περαιτέρω συζητήσεις ή κατά πόσον θα υπάρχουν ε, άλλες τέτοιες, ε, άλλα κείμενα. Όπως είπε και ο συνάδελφος μα πριν από λίγο, το θέμα είναι το εξής, ότι αυτό που προσπαθούμε να πετύχουμε δεν είναι σε καμία περίπτωση να ανακάμψουμε και να καθυστερήσουμε την συνένεση. Δεν σκοπεύουμε να κρατήσουμε το Τουρκμενιστάν εκτός της συμφωνίας σύνδεσης. Θέλουμε να πετύχουμε κάτι λογικό και μια επιτυχία σε ό,τι αφορά τις περαιτέρω εξελίξεις και προόδους και για το κράτος δικαίου και για το, τα, τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αυτό λοιπόν θεωρούμε ότι είναι ένας στόχος ε, εφικτός και ενδεχομένως να μας οδηγήσει και σε μια δραστηριότητα όπου θα θέλαμε να δούμε όλη την περιοχή να κινείται προς την κατεύθυνση αυτή, όχι μόνο του Τουρκμενιστάν και τις άλλες χώρες. Είναι σημαντικό ασφαλώς ε, παράγοντα και το Τουρκμενιστάν θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη. Ένα άλλο θέμα το οποίο δεν είχαμε συζητήσει κατά την συνάντηση, ένα πολιτικό ζήτημα. Η ομάδα μου εξετάζει το ενδεχόμενο Μάλλον αναρωτιέται ποια είναι η καλύτερη οδός να ε, συμμετάσχει η Επιτροπή της Βενετίας και οι συνταγματικές ε, μεταρρυθμίσεις, συνταγματικές αλλαγές που προτείνονται από πλευρά του Τουρκμενιστάν, ενδεχομένω να υπάρξει αξιολόγηση από την Επιτροπή της Βενετίας. Αυτό το απευθύνω ως ερώτημα, ως ζήτημα για την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, αλλά τονίζω και υπογραμμίζω ότι Συμφωνούμε απόλυτα με την εισηγητρία για την απόφαση και προτιθέμεθα ασφαλώ να συνεργαστούμε απόλυτα και στο μέλλον. Ευχαριστούμε πολύ. Ο Εντουάρτ έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δύο σύντομε παρατηρήσει επιτρέψτε μου να κάνω. Καταρχά, να ευχαριστήσω την εισηγητρία για τι προσπάθειε που έκανε να την ευχαριστήσω για τον δημιουργικό τρόπο με τον οποίο δεσμεύεται. Και πιστεύω ότι η θέση σε εφαρμογή της συμφωνίας με το Τουρκμενιστάν θα μπορούσε να αναπτύξει το πλήρες δυναμικό της χώρας και να δώσει πλήρη πλατφόρμα διαλόγου στην Ευρωπαϊκή Ένωση με τη χώρα αυτή. Και για να τονίσω αυτά που είπαν και οι προηγούμενοι ομιλητές. Τώρα είναι σημαντικό να συνεχίσουμε να δίνουμε πνοή στην πολιτική μας δέσμευση σε ό,τι αφορά τις σχέσεις με το Δουρκμενιστάν. Να μην επαναλάβουμε τα λάθη που κάναμε πριν από κάποια χρόνια, όταν ε, αφήσαμε αυτό το θέμα να περιπέσει σε χειμερία ανάρκη. Θα πρέπει να διοργανώσουμε αποστολή στη χώρα για να εκτιμηθεί η κατάσταση επιτόπου, να συνεχίσει η βελτίωση των, ε, να συνεχίσει να βελτιώνεται η επαφή με το Τουρκμενιστάν σε επίπεδο κόσμου και ανθρώπων. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Κούκαν και τώρα να δώσω τον λόγο στον επικεφαλής ε, της Εξυπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης για τις χώρες της περιοχής. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όπω ξέρετε, όπω ξέρουμε όλοι, οι διμερείς σχέσει μεταξύ του Τουρκμενιστάν και τη Ευρωπαϊκή Ένωση βασίζονται σε μια ενδιάμεση εμπορική συμφωνία από το 1998. Με άλλα λόγια, το τωρινό πλαίσιο για να συζητούμε πολιτικέ εξελίξει και ανθρώπινα δικαιώματα είναι πάρα πολύ περιορισμένο στι διμερεί μα σχέσει. Αυτό είναι ο λόγο για τον οποίο εμεί θα προτιμούσαμε να υπάρξει πρόοδο με την κύρωση μιας συμφωνία εταιρική σχέση και συνεργασία και θα μα δώσει το, ένα, σημαντικότερο, σημαντικό εργαλείο για να συζητήσουμε ευρύτερα θέματα. Να σας διαβεβαιώσω ότι συμμεριζόμαστε τις ανησυχίες σας για τα ανθρώπινα δικαιώματα στη χώρα αυτή και πάντα εγείρουμε τα θέματα αυτά των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε όλα τα επίπεδα. Αλλά μονάχα με μια τέτοια συμφωνία εταιρική και συνεργασίας θα υπάρξει ένα θεσμικό πλαίσιο και για τη συζήτηση αυτών των θεμάτων και θα επιτρέψει στην Ευρωπαϊκή Ένωση να προωθήσει περισσότερο τα θέματα αυτά η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και η ΥΠΑΤΗ έχουν ανταποκριθεί στην αίτηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να υπάρξει επιμερισμός πληροφοριών σε σχέση με την εφαρμογή ε, των σχέσεών μας σε επίπεδο ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Από πέρσι η Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης έχει κάνει περίπου 50 συναντήσεις με τη γραμματεία της ε, ΑΦΕΤ με τους ε, εισηγητέ και σχεδόν εισηγητέ όλα τα πολιτικά κόμματα για να του δώσουν πληροφορίες σε σχέση με την κατάσταση στο Τουρκμενιστάν. Είχαμε επίσης και διάσκεψη, με, με τηλεδιάσκεψη επαφή με πολλού κοινοβουλευτικού για τα θέματα αυτά. Έχουμε δώσει και μια έκθεση και στην Επιτροπή ε, Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ΤΡΟΑ, και θα κάνουμε το ίδιο και για το διάλογο του 2016 που έλαβε χώρα στις 17, Μαου 17 Μαΐου στις Βρυξέλλες. Και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει προσκληθεί σε συναντήσεις ε, <clears throat> με ε, την κοινωνία των πολιτών για τα θέματα αυτά. Επίσης θέλουμε να εξασφαλίσουμε ότι θα αντιμετωπιστούν τα θέματα των ατόμων που είναι αγνοούμενοι στο Τουρκμενιστάν όπως και σε άλλες χώρες. <clears throat> Θέλω λοιπόν να τονίσω ότι η Υπηρεσία Εξωτερική Δράση έχει προτείνει να υπάρξει και ανταλλαγή πληροφοριών για τα ανθρώπινα δικαιώματα στο Τουρκμενιστάν στα πλαίσια τη προετοιμασία μια νέα στρατηγική για τα θέματα αυτά. Αυτή η ανταλλαγή απόψεων επρόκειτο να λάβει χώρα μετά από την επίσκεψη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Τουρκμενιστάν που ήταν να γίνει τώρα, αυτό το μήνα, αλλά δυστυχώ αυτό το ταξίδι έχει ακυρωθεί. Μπορεί όμω να ξαναγίνει αυτή η ανταλλαγή απόψεων σε οποιαδήποτε ημερομηνία που είναι βολική για κάτι τέτοιο. Σε ό,τι αφορά τώρα αυτά τα οποία αναφέρθηκαν για τη χρήση τη επιτροπή τη Βενετίας και την εμπλοκή τη επιτροπή τη Βενετίας στην διαδικασία <clears throat> σύνταξη μιας, ενό νέου συντάγματο για το Τουρκμενιστάν, αυτό ήταν ένα θέμα το οποίο συζητήθηκε στον 8ο ετήσιο διάλογο ανθρωπίνων δικαιωμάτων με το Τουρκμενιστάν που είχαμε στι 17 Μαΐου στο Στι Βρυξέλλε, ο Υπουργό Εξωτερικών Χατζίεφ τόνισε ότι το Τουρκμενιστάν θα χαιρέτιζε θετικά οποιαδήποτε πρόταση οποιοδήποτε φορέα και οποιαδήποτε σχόλια για το σχέδιο συνταγματός τους. Για την δημιουργία μιας αντιπροσωπείας Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουμε τονίσει ότι εμείς συμφωνούμε απόλυτα με την αρχή ότι θα ήταν πολύ καλό να έχουμε μια πλήρη αντιπροσωπεία στο Τουρκμενιστάν αλλά προφανώς αυτό είναι θέμα και προϋπολογισμού και αυτό μέχρι στιγμή δεν έχει επιτρέψει στην υπηρεσία εξωτερική δράσης να έχει μια πλήρη αντιπροσωπεία στο Τουρκμενιστάν και παραμένουν από περιορισμοί ω προ τον προπολογισμό. <clears throat> Με την υποστήριξη βέβαια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μπορούμε να δημιουργήσουμε περισσότερε δυνατότητε προ την κατεύθυνση αυτή. Έχουμε στην Ασκαμπάντ ένα σύνδεσμο και ο πρεσβευτής μας στην Άγκυρα είναι επίσης αυτός ο οποίος ασχολείται πιο άμεσα με τα θέματα αυτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και τώρα θα δώσω το λόγο πάλι στην εισηγήτριά μας τη Ραμόνα Μανέσκο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους οι οποίοι πήραν το λόγο για να συμμετάσχουν σε αυτή τη συζήτηση. Πραγματικά συζητήσαμε λεπτομερώς ε, τη Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης και την ανάγκη να δοθεί συνένεση για αυτή τη συμφωνία, διότι, την PCA, διότι όπως είπαν οι συναδελφοί Κούκαν ε, και το Εύρο είναι το μόνο μέσο το οποίο μπορεί να είναι νομικά δεσμευτικό για τις αρχές του Τουρκμενιστάν. Θέλουμε λοιπόν να υποστηρίξουμε αυτή τη συγκατάθεση. Θέλω όμως ε, να πω ότι πολύ σωστά υπογράμμισαν και οι συναδελφοί μου σκιώδες ε, ότι υπάρχει ανάγκη για περισσότερες προσπάθειες από του Τουρκμενιστάν όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα, το κράτος δικαίου, τις ε, πραγματικές μεταρρυθμίσεις. Δεν θέλουμε λοιπόν να ανακόψουμε τη διαδικασία, ούτε να την κάνουμε να επαναχωρήσει. Θέλουμε απλά να βοηθήσουμε να δείξουμε ότι την υποστηρίζουμε πλήρως και ότι δεσμευόμαστε πολιτικά. Γι' αυτό το λόγο ε, καταλήξαμε σε αυτό το συμβιβασμό μιας ενδιέμεση έκθεσης βάσει του κανόνα 99, διότι θεωρούμε ότι αυτό θα διατηρήσει το ζήτημα εντός των συζητήσεων και προτεραιοτήτων μας. Θέλουμε δηλαδή να συνεχιστεί αυτό το έργο, διότι θέλουμε το συντομότερο δυνατόν να δώσουμε τη συγκατάθεσή μας για την PCA και έτσι να υποστηρίξουμε τις προσπάθειες της υπηρεσίας εξωτερικής δράσης για τη συνεργασία με το Τουρκμενιστάν. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ κυρία Μανέσκου. Μετά από τη συζήτηση αυτή είναι σαφές ότι θα προωθήσουμε το θέμα στο διευρυμένο Προεδρείο που θα αποφασίσει για τη συνέχιση της διαδικασίας ε, βάσει του αιτήματος της εισηγήτριας ε, συμπεριλαμβανομένης της προσωρινής αναστολής και του ανοίγματος της νέας διαδικασίας. Η γραμματεία μας ε, θα ενημερώνει την Επιτροπή. Ευχαριστώ πολύ για το σημείο 18 της ημερησίας διάταξης και περνάμε στο σημείο 19 της ημερησίας διάταξης αφορά τη στρατηγική ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως απάντηση στην προπαγάνδα από τρίτους εις βάρους της. Πρόκειται για μία έκθεση ίδιας πρωτοβουλίας, πολύ επίκαιρο θέμα, δεδομένης της τρέχουσας κατάστασης ε, όσον αφορά όλους τους τομείς πληροφοριών παγκοσμίω ε, και των διαδικτυακών χώρων. Η συγκήτρια είναι η κυρία Φωτίγκα από το ΙΣΕΑΡ, η οποία θα παρουσιάσει αναλυτικά την έκθεση αυτή. Εδώ θα γίνει η πρώτη ανταλλαγή απόψεων όσον αφορά τη στρατηγική ανακοίνωση ως απάντηση στην προπαγάνδα είναι ένα ζήτημα πολύ επικαιρό και πιστεύω θα μας βοηθήσει να αντιμετωπίσουμε το θέμα της παραπληροφόρησης των υβριδικών πληροφοριών προβλήματα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε ειδικότερα στο πλαίσιο της πολιτικής ε, ε, με την ανατολική σχέση όσον αφορά την επίθεση στην Ουκρανία, τη στάση της Ρωσίας, το πρόσφατο δημοψήφισμα στις κάτω ε, έχουμε μεγάλη παραπληροφόρηση Επίση και στο πλαίσιο της Συμφωνία Σύνδεσης Ευρωπαϊκής Ένωση Ουκρανίας πολλέ ε, λαθασμένες πληροφορίες κυκλοφόρησαν στο δημόσιο χώρο και χρειάζεται να παλέψουμε για να ε, λάμψει η αλήθεια και η πραγματική μα θέση. Για να είμαστε ισχυροί στη συζήτηση αυτή πρέπει να αναγνωρίσουμε, να κατανοήσουμε και να προσαρμοστούμε στι τακτικέ που χρησιμοποιούν οι αντίπαλοι μα. Ε, που παρουσιάζουν κάποιες ε, ειδήσει ως αληθείς, ε, έχουν ληφθεί ήδη σημαντικά μέτρα στο πλαίσιο της υπηρεσίας εξωτερικής δράσης, ειδικά τμήματα που ασχολούνται με την αντιμετώπιση της προπαγάνδας, αλλά θεωρώ ότι αυτό αποτελεί και μια πολύ καλή ευκαιρία για το Κοινοβούλιο να εκφράσει την άποψή του και τη θέση του, τη στάση του και τις συστάσεις του προ τα άλλα όργανα τη Ευρωπαϊκή Ένωση για το πώ θα μπορούσαμε να αντιμετωπίσουμε πιο αποτελεσματικά την προπαγάνδα και να προβάλλουμε αυτά που υποστηρίζουμε τις αξίες της ελευθερίας, της δημοκρατίας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του Κρατου δικαίου. Θα ήθελα λοιπόν να δώσω το λόγο στην κυρία Φωτίγκα, την εισηγήτρια. Έχετε το λόγο παρακαλώ. Αγαπητέ κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο. Συμφωνώ και επαυξάνω σε ό,τι αφορά αυτά που λέτε για τη σημασία των ζητημάτων ε, που συμφωνήθηκαν από το Προεδρείο σε ό,τι αφορά την έκθεση ίδιας πρωτοβουλίας. Επιτρέψτε μου να ευχαριστήσω καταρχάς Να ευχαριστήσω λοιπόν όλα τα εμπλεκόμενα μέλη, μέρη για την πρώτη αυτή έκδοχη της έκθεσης να ευχαριστήσω τη γραμματεία της ΑΦΕΤ, την κυρία Καμίνσκα, όλους και τους εκπροσώπους της Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης, την Δευθέντρια Σελβία Μοντζάτο, τον κύριο Πόρτσμαν, υπεύθυνο και αρμόδιο από ευρωπαϊκής πλευράς για την στρατηγική επικοινωνία της Ένωσης. Μία μικρή ομάδα που ξεκίνησε από τον κύριο Πόρτμαν σε ό,τι αφορά την καταπολέμηση της αρνητικής προπαγάνδας και της αρνητικής επικοινωνίας κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την επίθεση και την προσάρτηση ε, στην Κρυμαία. Και εκ των προτέρων και εκ των υστέρων. Θα ήθελα καταρχάς ε, να αναφερθώ στην φύση των απειλών που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αποτελεί μια μεγάλη απειλή και για πολλούς από εμάς ήταν και κάτι αναπάντεχο αυτό, η απειλή αυτή από την Ανατολή, από τη Ρωσική Ομοσπονδία, σε ό,τι αφορά τη στρατηγική επικοινωνία. Και ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την κρίση της Εσθονίας. Ύστερα υπήρχαν και άλλοι σημαντικοί παράγοντες. Σε ό,τι αφορά τα θέματα της γεωργίας, για παράδειγμα, και η επιχείρηση πρόσβαση σε κάποια τμήματα της γεωργίας και φυσικά η προσάρτηση της ε, Κρυμαίας. Αναγνωρίζονται λοιπόν αυτά από τους διεθνείς παράγοντες ε, της διεθνούς κοινότητας η απειλή που αντιμετωπίζουμε από τον Νότο, η αποσταθεροποίηση από τα Μαράκες μέχρι και τα Μπαγκλαδές και όλος ιδιαίτερος απειλές τρομοκρατίας. και από το εξωτερικό της άμεσης γειτονιάς μας και από την ίδια μας την επικράτεια, από διάφορες οργανώσεις όπως το Ισλαμικό κράτος. Η Αλκάιντα και άλλες οργανώσεις. Πολλές θα μπορούσα να αναφέρω. Η φύση δε της απειλής αυτής είναι τέτοια που αγγίζει όχι μόνο την ε, γειτονία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα σύνορα είναι τόσο θολά και ανάμεικτα που η επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα ίδια κρατημέλη είναι σε κίνδυνο. πρέπει να αντιληφθούμε, να περιγράψουμε και να κατανοήσουμε την πολυεπίπεδη αυτή απειλή σε ό,τι αφορά την στρατηγική επικοινωνία. Και σε πολλές περιπτώσεις να διευκρινίσουμε ότι σχεδιάζονται συγκεκριμένα για κάθε κράτος μέλος και για κάθε ενδεχόμενο στόχο της προπαγάνδας σε ό,τι αφορά την προπαγάνδα του Κρεμλίνου, της Ρωσίας. Γιατί πολλοί είναι αυτοί που διευκρίνησαν από τους κόλπους του Κοινοβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι θα προτιμούσαν το ρόλο του Κρεμλίνου. Ωστόσο, θα πρέπει να έχουμε αντίληψη του γεγονότος ότι σε ό,τι αφορά τη στρατηγική επικοινωνία, εκ παραλλήλου, αντιμετωπίζουμε παράλληλα και κρατικούς και μη κρατικούς φορείς σε ό,τι αφορά οργανώσεις όπως ε, η ΤΑΕΣ. Είναι σαφές ότι υπάρχει ένας ασύμετρος πόλεμος σε ό,τι αφορά την Ουκρανία έγιναν και κρατικές ε, απόπειρες υποστήριξης των υβριδικών αυτών προσπαθειών. Είναι εξαιρετικά πολύ σύμφωνο το θέμα αυτό και ήταν πάρα πολύ δύσκολο να διαρθρωθεί αυτή η έκθεση. Γιατί ακριβώς είναι τόσο καινοτομική η φύση του ζητήματος. Ωστόσο, χάρη στη συνεργασία και με τους κοιόδης εισηγητές, και με την βοήθεια του εκτελεστικού διευθυντή του κυρία Κουζανόφσκι καταφέραμε να παρουσιάσουμε αυτή την πρώτη εκδοχή του θέματος. Είναι εξαιρετικά πολύ σύμφωτο το θέμα. Και προκάλεσε ήδη σχόλια από το εξωτερικό. Αναφέρθηκε από το τεκτορικό Σπούτνικ και σχολιάστηκε. είναι περίεργο ότι ήταν, υπήρχαν ήδη εργαλεία για το ζήτημα αυτό το οποίο προσπαθούμε να περιγράψουμε. Αυτό σημαίνει ότι πραγματικά εφίσταται και είναι πραγματικά σημαντικό. Νομίζω δε ότι πολλοί πολιτικοί, ιδιαίτερα από τα παλαιά κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανέφεραν το πόσο τραυματική ήταν η είδηση ότι οι πολίτες των ίδιων τους των χωρών, νέοι άνθρωποι, θέλουν να συμμετάσχουν σε κάποιες από τις οργανώσεις αυτές. Είναι τεθειμένοι να ταξιδέψουν και να εκπαιδευτούν από το Ισλαμικό κράτος και στη συνέχεια να επιστρέψουν στην επικράτεια των κρατών μελών και να πολεμήσουν την ίδια τους την κοινωνία. Και πραγματικά αυτό αποτελεί μια τραυματική εμπειρία. Είναι περίεργο το πώς μπορούμε να κατανοήσουμε την φύση μιας τέτοιας απειλής. Πώς μπορούν να οριστούν τα εργαλεία, τα μέσα, οι τρόποι λειτουργίας και να αντιμετωπιστούν στη συνέχεια με όση επιτυχία είναι δυνατόν να σημειωθεί. Αυτό λοιπόν είναι κάτι το εξαιρετικά σημαντικό και θα ήθελα να αναγνωρίσω την τεράστια πρόοδο, το ορόσημο θα έλεγα, το οποίο σημείωσε η Λετωνική Προεδρία σε ό,τι αφορά το σκέλος αυτό. Εντοπίζοντας τα απαραίτητα μέτρα, τα οποία θα πρέπει να αναλυφθούν. Αναγνωρίζω ε, επίσης και χαιρετίζω το ανακοίνωση για τα κοινά μέτρα και τα κοινά σημεία του υπατού εκπροσώπου για τα ζητήματα αυτά. Είναι ένα θετικό βήμα και προσβλέπω στην ε, συμπερίληψη των σχολείων και παρατηρήσεων των σκιωδών εισηγητών. Ε, είμαι βέβαιη ότι θα είναι πολύ θετική η συνεργασία και αυτό το αντικείμενο πραγματικά αξίζει να εξευρεθεί μια συνένεση, μια πραγματική ουσιαστική συνένεση για μια πραγματική και ενδεχομένως καταστροφική απειλή για τα κάθε μελη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Φωτήκα και τώρα επειδή έχουμε πολλούς ομιλητές να περιοριστούμε σε 2-2,5 λεπτά για να μην ε, ξεπεράσουμε το χρόνο ομιλίας. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για τις εξαιρετικές της προσπάθειες. Και πιστεύω ότι ω αφετηρία θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τι αποφάσει και τι ανακοινώσει του Συμβουλίου και ειδικότερα τα συμπεράσματα του Μαρτίου 2015, καθώ ε, και την περιφερειακή στρατηγική τη Ευρωπαϊκή Ένωση για τη Συρία και το Ιράκ. Παράλληλα με αυτά, είναι σαφές ότι εδώ υπάρχει μια έλλειψη χρηματοδότησης. Επειδή ε, οι task βέβαια της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν κάνει καλή δουλειά, κάτι που πρέπει να λάβει υπόψη η έκθεση είναι η φύση της προπαγάνδας και της παραπληροφόρησης. Παραπληροφόρηση που έχουμε να αντιμετωπίσουμε όπως ε, το ότι ακριβώς δίπλα στα εξωτερικά σύνορα ε, ανατολικά και νότια της Ευρώπης ξεκινάει αυτή η παραπληροφόρηση, η οποία όμως καταλήγει στο κοινό της Ευρώπης. Κάτι άλλο που πρέπει να σημειωθεί είναι το ζήτημα της κοινή αντιμετώπισης ε, Ρωσίας και Ισλαμικού κράτους στο ίδιο έγγραφο, στην ίδια έκθεση. Θα έλεγα ότι εδώ έχουμε να κάνουμε με δύο όψεις του ίδιου νομίσματος, του ίδιου προβλήματος δηλαδή πληροφορίες που αποσκοπούν στο να αποδυναμώσουν δημοκρατικές αξίες, θεσμικά όργανα και συστηματική προπαγάνδα που οδηγεί σε ριζοσπαστικοποίηση και που καταστρέφει ζωές και τον ευρωπαϊκό τρόπο ζωής. Αυτή είναι η βασική προσέγγιση που θα αποτυπώνεται στις ε, τροπολογίες τις οποίες θα υποβάλω εγώ σύντομα. Φυσικά Προσβλέπω στη συνέχιση των εργασιών μα ε, για την εκθέση αυτή μαζί με την κυρία Φωτίγα και του λοιπού συναδέλφου σα. Ευχαριστώ πολύ. Αυτά είχα να πω προ στιγμή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Ούγγουρε Ο κύριο Φρόιντ έχει το λόγο, ο οποίο είναι σκιώδη συζητητέ από τη Σοσιαλιστική Ομάδα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Την κυρία Φωτίγκα, πού είναι για την πάρα πολύ καλά δομημένη αυτή έκθεση για το πώς θα αντιμετωπίσουμε την προπαγάνδα και την παραπληροφόρηση η οποία κατευθύνεται κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προτού όμως οι λεπτομέρειες του σχεδίου έκθεσης να πω ότι θα πρέπει να δούμε αν μπορούμε να βρούμε μια κοινή γλώσσα, ένα κοινό ορισμό της προπαγάνδας. Όπως ξέρουμε, ξεκινώντας από το 1930 με το ναζιστικό καθεστώς, ένα ειδικό γραφείο, ακόμα και μια κυβερνητική θέση, δημιουργήθηκε το Propaganda Ministerium ώστε να διαχέει πληροφορίες που οι Ναζίδες θέλαν να ε, χρησιμοποιήσουν. Και οι Ναζί χρησιμοποίησαν ακριβώς την έννοια της προπαγάνδας, γιατί θέλαν να διαχέουν ιδέες, ε, φήμες, ψευδείς ειδήσει οι οποίες θέλαν με τον τρόπο αυτό να επηρεάσουν και να χειραγωγήσουν την κοινή γνώμη. Οι Δύση και ιδίω οι Ηνωμένε Πολιτείε δεν αδράνησαν, δημιούργησαν τα δικά του εργαλεία, αντιμετωπίζοντα καταρχήν την προπαγάνδα των Ναζί και μετά την σοβιετική ε, προπαγάνδα που ήταν προφανώς μορμερής. Εργαλεία όπως η Φωνή της Αμερικής, που υποστηρίχθηκαν βέβαια από το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ, χρησιμοποίησαν τη συλλογή πληροφοριών τους στις δυτικές δημοκρατίες, προσπαθώντας να μεταλαμβαδεύσουν τις δυτικές αξίες σε χώρες όπου η πληροφορία ήταν απόλυτα υποέλεγχο. Οι ιστορικοί αναγνωρίζουν σήμερα ότι στη συνέχεια οι, δικοί, οι δορυφόροι επικοινωνιών που επέτρεψαν να εκπέμπονται προγράμματα πέραν των χωρών παραγωγής τους συνέβαλαν στην πτώση του σιδηρού παραπετάσματος και των κομμουνιστικών καθεστώτων. Για το σχέδιο έκθεση τώρα θα ήθελα να εκφράσω κάποιες επιφυλάξεις. Και δεν συμφωνώ να αναμειχνύεται στην ίδια έκθεση η προπαγάνδα του Νταέσ και της Ρωσίας στην ίδια έκθεση. Ο δυτικός πολιτισμός νομίζω ότι συμφωνεί ότι το Ισλαμικό κράτος ή το Νταέσ δεν είναι κράτος αντίθετα με τη Ρωσία το να αναγάγουμε τον ΤΑΕΣ σε επίπεδο κρατικής ενότητας και να θέσουμε τους δύο αυτούς τις δύο αυτές οντότητες, τη Ρωσία και τον ΤΑΕΣ, στην διέκθεση είναι κάπως αντιπαραγωγικό κατά την άποψή μου. Τούτου λεχθέντος. Δεν χωρεί αμφιβολία ότι σε διάφορα τμήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης η ρωσική προπαγάνδα αντιμετωπίζεται με διαφορετικό τρόπο. Η Πολωνία μπορεί παραγωγικά να υφίσταται ένα μεγαλύτερο μπαράζ απόψεων που υποστηρίζουν το Κρεμλίνο από την Πορτογαλία. Πρέπει να βρούμε λοιπόν μια κοινή γνώμη η οποία να εφαρμόζεται σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι μοναχά στις χώρες που είναι όμορες της Ρωσίας. Και δεύτερον, πιστεύω είναι σημαντικό να κάνουμε μια διάκριση μεταξύ της κακής προπαγάνδας και της καλής πληροφόρησης. Πολύ συχνά πρέπει να χρησιμοποιήσουμε συγκεκριμένα εργαλεία για να δούμε σε ποιο βαθμό μια προπαγάνδα πράγματι φτάνει στην κοινή γνώμη και επηρεάζει ένα σημαντικό αριθμό ατόμων. Αυτή τη στιγμή δεν ξέρουμε πώς οι άνθρωποι παρακολουθούν ή ακούν ε, τηλεοπτικά προγράμματα ή ραδιοφωνικά προγράμματα που είναι φιλικά προς το Κρεμλίνο και επηρεάζονται από αυτά. Ίσως η προπαγάνδα αυτή που δεν αμφιβάλλω ότι υπάρχει, ίσως αυτή η προπαγάνδα ε, αυτή τη στιγμή Προφανώ φτάνει στι χώρε μα, αλλά δεν υπάρχει, κάποιο, δεν υπάρχει πολλοί κόσμο ο οποίο είναι κολλημένο στην τηλεόραση και παρακολουθεί την προπαγάνδα τη Ρωσία. Και κάτι ακόμα λοιπόν, δεν θέλω να προτρέξω των γεγονότων, ούτε να απορρίψω αυτή την πρόταση. Θα ήθελα να έχω περισσότερε λεπτομέρειε προτού ξεκινήσουμε να αντιμετωπίσουμε και να αναχαιτήσουμε κάτι το οποίο μπορεί, αλλά μπορεί και όχι, να είναι μια σημαντική απειλή για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο κύριο Αουστρεβίτσιου έχει το λόγο από την άλλη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όπως γνωρίζουμε όλοι, τα ψέματα που επαναλαμβάνονται πολλές φορές αρχίζουν να μοιάζουν με αλήθειες. Και αν παραβλέψουμε αυτό το πρόβλημα και την πραγματικότητα, μπαίνουμε μέσα σε νέες παγίδες. Όλοι μας είμαστε μάρτυρες ενός υβριδικού πολέμου. Αυτό είναι αδιαμφισβήτητο. Αποτελεί κομμάτι της πραγματικότητας. Ένα από τα πιο αποτελεσματικά μέσα υβριδικού πολέμου, ειδικότερα στα πρώτα στάδια, είναι η προπαγάνδα. Η προπαγάνδα που στοχεύει συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες, ε, περιοχές, χώρες, λαούς. Πρέπει να παραδεχτώ ότι αυτή η έκθεση ιδίας πρωτοβουλίας ε, της ε, συναδέλφου Φορτίγα βασίζεται σε αδιαμφισβήτητα θεμέλια. Πρέπει, πιστεύω, ε, υπάρχουν αρκετά σωστή λόγια να υιοθετήσουμε αυτή την έκθεση, αλλά θα πρέπει να κάνουμε κάποιες προτάσεις από πλευράς μας για να προωθήσουμε και τις δικές μας απόψεις, τι πιστεύουμε Εμεί, Παρ' όλα αυτά πρόκειται για ένα καλό έγγραφο, ένα καλό σχέδιο για το... τις που θα πρέπει να κάνουμε εμείς. Πράγματι, συνάδελφοι, η προπαγάνδα δεν γνωρίζει σύνορα. Για να το πω διαφορετικά, δεν παραδέχονται όλοι οι ασθενείς ότι έχουν μολυνθεί. Λένε οι συναδέλφοι ότι κάποιε χώρε δίπλα στη Ρωσία, ο λέει ότι κάποιε χώρε δίπλα στη Ρωσία ίσω έχουν μολυνθεί περισσότερο από την προπαγάνδα. Ε, η Γερμανία, ο γερμανικός λαός χρειάστηκε να περάσει, να ζει στην ιστορία της Λίζα ενός κοριτσιού που κατασκευάστηκε από τη Ρωσία για να αναγνωρίσει σε ποιο βαθμό η χειραγώγηση της κοινή γνώμης αποτελεί πλέον τακτική της Μόσχας. Και αυτό δεν είναι παρά μόνο ένα παράδειγμα. Ας μην υποτιμάμε λοιπόν ούτε να είμαστε υπεραισιόδοξοι όσον αφορά τις ζημιές που προκαλεί η προπαγάνδα. το μέγεθος της χώρας ε, έχει ελάχιστη σημασία μάλιστα. Ε, για την έκθεση αυτή θα ήθελα να υπογραμμίσουμε περισσότερο την πολύ απαραίτητη συνεργασία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΝΑΤΟ μπορεί να φέρει πολύ καλά αποτελέσματα. Το ΝΑΤΟ είναι ένας, μια αμυντική συμμαχία ε, με δυτικές αξίες που υποστηρίζει τον δυτικό τρόπο ζωής. Οι στόχοι μας είναι παρεμφερείς, παρότι χρησιμοποιούμε διαφορετικά μέσα. Γι' αυτό λοιπόν η συνεργασία αυτή πιστεύω δεν επιδέχεται αμφισβήτηση. Τώρα, οι δραστηριότητες που σχετίζονται με προπαγάνδα που προέρχεται από εχθρικές ε, χώρες θα πρέπει να αντισταθμιστούν μέσα που θα χρησιμοποιηθούν εδώ στη κράτη-μέλη μας και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πιστεύω ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει να έχουν ως γραμμή πολιτική στο να βελτιώσουν τις ικανότητέ του, ανάλυση των πληροφοριών και λήψη των απαραίτητων αποφάσεων όσον αφορά ε, εχθρικέ ε, πληροφορίες ε, και τα προληπτικά μέτρα που θα πρέπει να υιοθετηθούν. Τέλος, θα ήθελα να υπογραμμίσουμε λίγο περισσότερο τη γειτονία. Επειδή αναγκαζόμαστε να συνεργαστούμε με χώρες οι οποίες επηρεάζονται και μολύνονται σε μεγάλο βαθμό από τις εχθρικές αυτές πληροφορίες στη γειτονία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό αποτελεί ήδη κομμάτι της πολιτικής γειτονίας μας και αφορά ορισμένους γειτονές μας ε, να υπάρξει λοιπόν πιο αποτελεσματική συνεργασία μέσω κοινών προγραμμάτων και ανταλλαγή πληροφοριών. Για να ολοκληρώσω τα συγχαρητήριά μου στη συνάδελφο, η οποία κατέβαλε εκπληκτικές προσπάθειες ε, για την προσέγγιση ε, αυτού του θέματος σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και ελπίζουμε ότι, ελπίζω ότι αυτή η εκθέση δεν θα είναι το τελευταίο βήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως αντίδραση και ως δράση, δράση μάλλον χωρίς να είναι άμεση αντίδραση σε αυτή την προπαγάνδα και για την αντιμετώπιση της. Ευχαριστούμε. Κύριε Χάνης, παρακαλώ. Και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Φωτίγκα για το πνεύμα συνεργασίας και την, ε, ε, να ευχαριστήσω την κυρία Μοκερίνιο και τους ε, υπαλλήλους της ε, Stratcom, γιατί ουσιαστικά βρισκόμαστε ένα βήμα παραπέρα. Εσείς μάλλον βρίσκεστε ένα βήμα παραπέρα από ότι βρισκόμαστε εμείς σε ό,τι αφορά το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Δημοκρατία και έτσι κάναμε ένα πρώτο βήμα για το πώς θα αντιμετωπίσουμε μια νέα κατάσταση σε ό,τι αφορά την προπαγάνδα που στρέφεται κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης Θεωρώ ότι ο συνάδελφος κ. Φρόιντ έθεσε κάτι πάλι σημαντικό. Έχουμε στην Ήπειρο μας εμπειρία με την προπαγάνδα, προπαγάνδα με κακό σκοπό. Αλλά ακριβώς επειδή έχουμε συλλέξει πολλές εμπειρίες, θα πρέπει πλέον να είμαστε πιο σόφρονες σε μια νέα κατάσταση η οποία αποκρισταλώνεται και στην οποία καλούμαστε να αντιδράσουμε με πιο σόφρονα τρόπο. σε ό,τι αφορά την προπαγάνδα του Ισλαμικού κράτους και του ΙΣΙΣ, θεωρώ ότι θα πρέπει να καταταχθούν με διαφορετικό τρόπο σε σχέση με την απειλή που αποτελεί για μας το Κρεμλίνο. Και νομίζω ότι η προπαγάνδα του Κρεμλίνου συνειδητά στρέφεται κατά της σταθερότητας και της ομόνοιας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αντίθετα με εσά, κύριε Φρόιντ, δεν πιστεύω ότι σε πρώτη γραμμή στρέφεται κατά των Ανατολικό Ευρωπαίων, αλλά ότι εδώ και καιρό στο στόχαστρο βρίσκεται ο στόχος του να ειδωθεί η Ρωσία με διαφορετικό τρόπο από ό,τι είναι στην πραγματικότητα και ο, δίος, ο ίδιος ο Πούτιν ε, προβλήθηκε ως υποστρακτής και μάλλον θαυμαστής του, μάλλον θαυμαστής του Κόμπελ, το οποίο μου προκάλεσε πραγματικά φρίκη. Και νομίζω ότι είναι και οι Ρώσοι πολίτες εκείνοι που πλήττονται από την ε, νέα αντιμετώπιση της προπαγάνδας αυτής. Και πιστεύω ότι το πρώτο πράγμα που είναι απαραίτητο είναι να ε, εντοπίσουμε το τι αποτελεί προπαγάνδα. Να μπορεί ο πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης να είναι σε θέση να αναγνωρίζει καν την προπαγάνδα και ότι αυτό αποτελεί κάτι το επικίνδυνο και ότι ε, διακυβεύει το δημοκρατικό μας σύστημα. Η συστηματική λοιπόν σύνδεση της προπαγάνδας ε, που έχει πάρα πολύ καλή χρηματοδότηση. και ε, η συστηματική σύνδεση με την υποστήριξη ακροδεξιών, εξτρεμιστικών, ε, αντιευρωπαϊκών κινημάτων. Αυτό πραγματικά θα πρέπει να θεωρήσουμε πολύ επικίνδυνο. Και πώς αντιδρούμε λοιπόν στα ψέματα, στις θεωρίες, συνωμοσίες, στις μισοαλήθειες, σε στρατηγικές ε, που κάνουν τον κόσμο να φοβάται, στρατηγικές ε, της Δούμας. Με την απόπειρα να ενημερώσουμε σωστά με τις ε, προσπάθειες της καλής δημοσιογραφίας. Αυτά τα συζητήσαμε και χθε και νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να πραγματοποιήσει το ρόλο αυτό, αλλά πρέπει να το θέλει κιόλας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε Κυρία Χάραμς. Στέτινα, please. Ο κύριος Στέτινα έχει το λόγο τώρα. Χωρίς μικρόφωνο μιλητής. Ναι, ναι, συγγνώμη. Ξαναρχίζω. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Φωτίγα γιατί είναι ένα βασικό ενιολογικό σχέδιο αυτό το οποίο παρουσιάζει η έκθεσή της. Είναι σημαντικό ότι η έκθεση αυτή ασχολείται με τα θέματα της Ρωσίας. Είναι κάτι το οποίο ελέγχθη ότι η Ρωσία διεξάγει ένα υβριδικό πόλεμο κατά χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά εναντί ποιανού στρέφεται αυτός ο υβριδικός πόλεμος. Εναντί ποιου γίνεται αυτή η προπαγάνδα ψευδών. Εγώ πιστεύω ότι έχει μονάχα ένα στόχο και αυτός είναι να εξολοθρεύσει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι λοιπόν μια πιο επικίνδυνη και αποτελεσματική από ό,τι πυραυλικά συστήματα ή άρματα μάχης. Και ο στόχος λοιπόν είναι σαφής και αυτό αναφέρεται και στην έκθεση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν δεν αντιμετωπίζει παρά μόνο ασθενικά αυτά τα πάρα πολύ αποτελεσματικά όπλα του Κρεμλίνου. Γνωρίζετε όλοι ότι η κυρία Μογκερίνη πρόσφατα ε, έχει πάρει την εντολή από το Συμβούλιο να δημιουργήσει μία ομάδα η οποία θα αντιμετωπίσει την προπαγάνδα που προέρχεται από τη ρωσική κυβέρνηση. Και αυτή η ομάδα έχει οκτώ μέλη. Μα μπορείτε εσείς να αντιμετωπίσετε μια εξατία εκατομμυρίων που εκπορεύεται από το Russia Today και από τους Σπούτνικ και από άλλα εργαλεία προπαγάνδας της ρωσικής προπαγάνδας που δημιουργούν και διοχετεύουν τόσα πολλά ψέματα. Δεν μπορεί λοιπόν να γίνει κάτι τέτοιο. Εμείς θα πρέπει, όπως τονίζεται και στην έκθεση, θα πρέπει να ασχοληθούμε με το θέμα της χρηματοδότησης, της αντιμετώπισης αυτής της ε, προπαγάνδας. Δεν θέλουμε εμεί να χάσουμε αυτό τον πόλεμο τη πληροφορία και δεν μπορούμε να τον κερδίσουμε αν δεν χρησιμοποιήσουμε τα απαραίτητα κονδύλια. Ευχαριστώ. Ο κύριο Μάμικιν έχει τώρα το λόγο. Ε, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα, αγαπητοί συνάδελφοι, να θέσω το εξή ερώτημα. Βλέπετε συχνά τα μέσα ενημέρωσης που αναφέρονται στο σχέδιο έκθεσης, τα ρωσικά αυτά μέσα που αναφέρονται και αν τα, τα παρακολουθείτε, σας έχουν επηρεάσει, σας έχουν οδηγήσει σε αλλαγή άποψης. Μιλάμε για κάποιες ομάδες του πληθυσμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση που βλέπουν αυτά τα μέσα ενημέρωσης ή διαβάζουν τις αντίστοιχες εφημερίδες. Ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι, τι ξέρουμε για αυτούς, σε ποιες χώρες είναι, δεν λέει τίποτα η έκθεση όλα αυτά, ποια είναι η μητρική του γλώσσα. Εγώ ξέρω μονάχα μια τέτοια ομάδα στην Λετωνία. Περίπου 15% του πληθυσμού της Ρωσίας είναι ουσιαστικά αλλοδαπή επίσημα. Ε, είναι πρώην Ρώσοι πολίτε. Δεν έχουν καμία όμω υπηκότητα ούτε λετονική ούτε τίποτα άλλο. Δεν μπορούν να ψηφίσουν ούτε για τοπικέ ούτε για βουλευτικές εκλογές. 25 χρόνια είναι απόκληροι από την εκλογική διαδικασία. Τι μπορούμε να πούμε λοιπόν για τη λειτουργία τη δημοκρατία. Θα πρέπει να θέσουμε λοιπόν αυτό το ερώτημα. Γιατί υπάρχει ένα τόσο μεγάλο μέρο του πληθυσμού τη Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν μπορεί να ψηφίσει ούτε καν σε τοπικέ εκλογέ. Αυτό δεν είναι προπαγάνδα του Πούτιν. Είναι ένα πραγματικό πρόβλημα το οποίο δεν έχει λυθεί εδώ και 25 χρόνια. <clears throat> ένα τέταρτο αιώνα. Γι' αυτό έχουν μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στα μέσα ενημέρωση τη Ρωσία από ότι στη δικιά του κυβέρνηση. Και αυτό το παράδειγμα δείχνει ότι πρέπει να εστιάσουμε όχι σε ένα αφηρημένο αγώνα προπαγάνδας, αλλά στο να λύσουμε τα πραγματικά προβλήματα των πολιτών μας. Ευχαριστώ. Ο κύριος Γιούρεκ έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα κυρίως να ευχαριστήσω την κυρία Φώτικα για την εξαιρετική αυτή πρωτοβουλία και για το γεγονός ότι πραγματικά υπέδειξε ότι θα πρέπει να αναρωτηθούμε για τα ζητήματα αυτά για το πώς θα πρέπει να προσπίσουμε τα συμφέροντά μας. Και θα ήθελα μόνο αναφερθώ στο εξή. Γίνεται αναφορά και θα έπρεπε να γίνεται αναφορά στην έκθεση σε δύο ζητήματα. Καταρχά, στο γεγονό ότι θα πρέπει να θυμόμαστε ότι οι σημερινέ ρωσικέ αρχέ προσπαθούν μεν να κρύψουν την προπαγάνδα τους, αλλά συνολικά έχουν μια γεωπολιτική κατεύθυνση η οποία συνεχίζει στην παράδοση της Σοβιετικής Ένωσης και πρόκειται για ένα θέμα κοινωνικής ανισότητας. Ένα μεγάλο τμήμα της κοινωνίας δεν μπορούσε να συμμετέχει στα κόμματα, στους εσωτερούς κύκλους, αν θέλετε, των κομμάτων. Δεν ε, πρόκειται λοιπόν για μια ε, εποχή χειραφέτησης της πλειοψηφίας όπως ε, παρουσιάζεται. Θα πρέπει λοιπόν να αναφέρουμε ακριβώς το μεγάλο τμήμα αυτό της κοινωνίας. Αυτός ο νέος καπιταλισμός λοιπόν ουσιαστικά αποτελεί μια κατ' ουσίαν συνέχιση της Ιωβετικής Ένωσης, της Ολιγαρχίας. Παράλληλα υπάρχει και μια προπαγάνδα κατά της Δύσης. Ε, στο σημείο αυτό θα πρέπει να αντιληφθούμε το τι υποστηρίζουν και η έκθεση θα πρέπει να αναφέρει το γεγονός ότι εμείς εκπροσωπούμε ιστορικές αξίες, ε, ιστορικές ιδέες των χωρών μας. Η προπαγάνδα διαμορφώνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να εκμεταλλεύεται κάθε μεμονωμένο στοιχείο της πολιτικής μας. Αλλά Βιετνάμ, Κούβα, ούτω καθεξής, όλες αυτές οι κοινωνικές ε, συνθήκες, όλα αυτά τα κοινωνικά στοιχεία έχουν συμπεριληφθεί στην προπαγάνδα και αυτό αποτελεί προφανώς την ιδεολογία του Λέιν και θα πρέπει στο σημείο αυτό να ξεκαθαρίσουμε ότι εμείς θέλουμε να υπερασπιστούμε τις αξίες των ιστορικών μας εθνών. Προασπιζόμαστε τη Δύση που είναι σε θέση να εγγυηθεί την εξαρτησία των κρατών και δεν θέλουμε να εφαρμοστεί αυτή η πολιτισμική κρίση που προκύπτει από την Σοβιετική Ένωση. Υπάρχουν λοιπόν διάφορα στοιχεία τα οποία τα βλέπουμε, τα ανταλαμβανόμαστε, αλλά δεν τα υποστηρίζουμε. Σα ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρο. Ευχαριστούμε τον συνάδελφο Γιούρεκ και τώρα να δώσω το λόγο στον συνάδελφο Στρογεύσκη, ο οποίο προετοιμάζει μια γνωμοδότηση από πλευρά τη Επιτροπή Πολιτισμού για το ζήτημα αυτό. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, πρώτα απ' όλα, εδώ έχουμε μια πάρα πολύ σημαντική έκθεση, ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα και προφανώς είναι και σημαντικό πρόβλημα. Δεν μπορούμε λοιπόν σε καμία περίπτωση να παραγνωρίσουμε το ζήτημα αυτό. Και έρχεται και καθυστερημένα η αντίδρασή μας νομίζω σε αυτή την προπαγάνδα η οποία έχει λάβει μεγάλες διαστάσεις. Θέλω να υπογραμμίσω τα εξή. Αυτή τη στιγμή η Ευρώπη δεν έχει καμία άμυνα εναντίον αυτής της προπαγάνδας. Δεν έχει τα απαραίτητα εργαλεία για να αντιμετωπίσει αυτή την προπαγάνδα. Δεν υπάρχει κανένα μέσο για την αντιμετώπιση και δεν υπάρχουν και προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης ώστε οι νέοι στα σχολεία να εμποδιστούν από το να επηρεαστούν από την προπαγάνδα αυτή. Και οι νέοι δεν μαθαίνουν να ξεχωρίζουν το πολιτικό μάρκετινγκ από την προπαγάνδα. Νομίζω λοιπόν ότι είναι φανερό ότι υπάρχει μια προπαγάνδα η οποία έχει όλο και μεγαλύτερη επιρροή στην κοινή γνώμη και έχει σαν στόχο να κατακτήσει την κοινή γνώμη και να την ε, κατακτήσει με στοιχεία τα οποία είναι ψευδή. Ξέρουμε όλοι όμως η προπαγάνδα δεν έχει καμιά σχέση με την πληροφόρηση. Πρέπει λοιπόν να αντιμετωπίσουμε την παραπληροφόρηση, τις ε, μονομερείς και μερικές πληροφορήσεις και την λανθασμένη ερμηνεία της πραγματικότητας. Ό,τι δεν έχει να κάνει με την πραγματικότητα θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε μαζί με την προπαγάνδα. Όλα αυτά τα πράγματα είναι απαραίτητα, είναι απολύτως απαραίτητα εμείς να πούμε ότι η προπαγάνδα είναι κάτι που προέρχεται από μια χώρα, μια περιοχή. Όχι, είναι ένα συνολικό φαινόμενο και μέσα στο πλαίσιο αυτό η Ευρώπη απειλείται από την προπαγάνδα. Είναι πολύ σημαντικό και το λέω κλείνοντας. Φαίνεται ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας υβριδικός πόλεμος ο οποίος έχει ξεκινήσει εναντίον μας και θα πρέπει και σε σχέση με αυτόν τον πόλεμο να αναπτύξουμε τα κατάλληλα εργαλεία. Δεν φτάνουν τα συμβατικά όπλα για ένα τέτοιο πόλεμο. Πρέπει να υποστηρίξουμε τις αρχές μας χρησιμοποιώντας και εμείς υβριδικά όπλα, τεχνολογική καινοτομία, ώστε να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε στεναρά την προπαγάνδα εναντίον μας και να εμποδίσουμε ότι θα επηρεάσουν τους ανθρώπους στην κοινωνία μας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό με αυτές τις δραστηριότητες να μην απαντήσουμε με δική μας προπαγάνδα. Οι ευρωπαϊκές αρχές όμως είναι αρχές που δεν αποτελούν προπαγάνδα, θα πρέπει να, να διακριθούν από την προπαγάνδα και να τονιστεί ότι είναι κάτι διαφορετικό. Θέλουμε Ξέρω λοιπόν ότι είναι η πρόθεση των συντακτών της έκθεσης να αντιμετωπίσουν την προπαγάνδα. Εμείς όμως θα πρέπει να αντιπαραθέσουμε στην προπαγάνδα τις πραγματικές αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ώστε να είναι οπλισμένοι με αυτές και να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν την προπαγάνδα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ο Αντώνιο Ευχαριστώ Πρόεδρε, πολύ σύντομα. Επειδή ακόμα βρισκόμαστε σε φάση ανταλλαγής απόψεων, ήθελα να σας αναφέρω κάποιους προβληματισμούς μου όσον αφορά τις εργασίες αυτές που είναι μεν πολύ σημαντικές. Αλλά πρώτα απ' όλα υπάρχουν κάποιοι κίνδυνοι που θα πρέπει να αποφύγουμε. Όπως ε, η στρεβλωμένη άποψη ε, για μια συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή όπως η Ρωσία τι, το, ο κίνδυνος που να με τη Ρωσία με τον ΤΑΕΣ. Ε, θα πρέπει να μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά μεταξύ των δύο αυτών. Διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος ε, να διαπράξουμε ένα πολιτικό λάθος σοβαρότατο. Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι χρειάζεται να εμβαθύνουμε περισσότερο τα τεχνικά μέσα και τους χειρισμούς που θα πρέπει να γίνουν όχι μόνο στον τομέα της πληροφορικής αλλά και γενικότερα. Όχι μόνο για να παρακολουθούμε καλύτερα την κατάσταση αλλά και για να έχουμε πιο καλά συντονισμένες δράσεις που να αντιμετωπίσουν την ε, προπαγάνδα αυτή ειδικότερα χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα εργαλεία. Θα πρέπει λοιπόν να προσπαθήσουμε να προσδιορίσουμε τα σωστά εργαλεία ώστε η Ευρώπη μέσω της επένδυσης που θα κάνει να ανταποκριθεί σωστά. Το τρίτο που θα ήθελα να πω Ωραία, παραδεχόμαστε ότι η προπαγάνδα αυτή είναι μια από τις ισχυρότερες ε, ε, ότι συγγνώμη, η ισχυρότερη προπαγάνδα κατά της Ευρώπης προέρχεται από την ίδιες χώρες της Ευρώπης αλλά σε αυτό το έγγραφο θα πρέπει να εμβαθύνουμε περισσότερο και την πολιτική απόκριση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, όσον αφορά την προπαγάνδα που έρχεται από τρίτου. Είναι κάτι που έχουμε συζητήσει πολλέ φορέ στο θέμα των αξιών, αλλά εγώ πιστεύω ότι ε, τίθεται κυρίω το ζήτημα τη ευρωπαϊκή ταυτότητα. Διότι όταν ε, κλονίζεται αυτή η ταυτότητα από εξωτερικού παράγοντε, είναι πολύ εύθραστοι και πιο ευάλωτη σε αυτούς τους εξωτερικού παράγοντε. Εάν ε, αποφύγουμε αυτό το θέμα, θα αποτελούμε όλο και μεγαλύτερα θύματα των τέτοιων εξωτερικών επιδρομών. Ε, είναι ένα θέμα το οποίο δεν μπορούμε να αποφύγουμε, πρέπει να το συζητήσουμε. Ε, γιατί υπάρχει αυτός ο κίνδυνος αποσύνθεσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, βρισκόμαστε σε μια πολιτική διαδικασία και καθόμαστε και συζητάμε για μια προπαγάνδα άλλων, ενώ εμείς καταστρεφόμαστε, καταστρέφουμε εμείς οι ίδιοι τον εαυτό μας. Αυτά τα δύο στοιχεία είναι πολύ σημαντικά και πρέπει να τα εξετάσουμε ταυτόχρονα, την πολιτική πτυχή με την ανάγκη φυσικά να αντιμετωπίσουμε και τις εξωτερικές επιθέσει. Αυτό λείπει πιστεύω από την έκθεση. Πολύ ενδιαφέρουσα η πρότασή σας. αν ακολουθήσουμε αυτά που λέει ο κ. Φρόιντ θα βάλουμε στην άκρη τον ΤΑΕΣ ε, και θα συμπεριλάβουμε την ε, ευρωπαϊκή ταυτότητα, αλλά αυτό αλλάζει λίγο το σκεπτικό της έκθεσής μας. Ε, δίνω τώρα το λόγο στον κύριο Πιτίδιο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, στην έκθεση του ψηφίσματος για την αντιμετώπιση της προπαγάνδας των τρίτων κατά της Ευρωπαϊκής Ενώσεως περιλαμβάνεται και η Ρωσία. Αυτό κατά την άποψή μου είναι αντιφατικό σχετικά με την πολιτική που εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Απ' τη μια μεριά θεωρούμε τη Ρωσία ως στρατηγικό εταίρο, συνεργαζόμαστε μαζί της, κάνουμε συμφωνίες για το πώς θα αντιμετωπίσουμε την κρίση της Συρίας και απ' την άλλη πλευρά ερχόμαστε να θεωρήσουμε την Ρωσία εχθρική χώρα. Διότι ως γνωστόν η προπαγάνδα είναι μια ενέργεια η οποία εκτοξεύεται από μια εχθρική χώρα προς άλλη εχθρική χώρα. Άρα λοιπόν πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τι ακριβώς θέλουμε. Θεωρούμε τη Ρωσία εχθρική ή όχι. Αν θεωρούμε εχθρική, ναι, τότε να δούμε ποια είναι η προπαγάνδα τη και να την αντιμετωπίσουμε. Εάν όμως θέλουμε να την έχουμε εταίρο στρατηγικό, τότε πρέπει να πάψουμε να τη θεωρούμε εχθρική, αλλά δεν πρέπει να μιλάμε για προπαγάνδα ρωσική. Άλλωστε, στη σημερινή εποχή, η έννοια της προπαγάνδας και τη ενημερώσεω έχει ε, πολύ διασταλεί. Δηλαδή, δεν ξέρει κανεί ποια είναι η ενημέρωση, ποια είναι η προπαγάνδα. Εκείνο το οποίο πρέπει να γίνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι το να λέμε την αλήθεια, διότι μία από τι αρχέ τη προπαγάνδα είναι να υπάρχει συνάφεια μεταξύ των όσων λέγονται και των όσων πραγματικά συμβαίνουν. Δεν μπορούμε να λέμε, παραδείγματο χάρη, γιατί δεν γινόμαστε αξιόπιστοι, ότι μεταξύ των χωρών της Ευρώπης υπάρχει αλληλεγγύη και να έχουμε επί έξι χρόνια την Ελλάδα σε μια κατάσταση απαράδεκτης οικονομικής εξαθλιώσεως και μετά να θέλουμε να γίνουμε αξιόπιστοι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πολύ σημαντική και πολύ καλή. Επιπλέον, εάν θέλουμε να γίνουμε πραγματικά αποδεκτοί από τις κοινωνίες μας, πρέπει να διορθώσουμε τα λάθη μας και να προχωρήσουμε. Και τελειώνω κάνοντας τρία, απευθύνοντας συγγνώμη τρεις ερωτήσεις προς την ε, κυρία Φόντικα που ε, έγραψε αυτή την ενδιαφέρουσα έκθεση αναφέρει σε κάποια στιγμή ότι η Ρωσία χρησιμοποιεί ως μέσον προπαγάνδας την Ορθόδοξη Εκκλησία. Επειδή ω Έλληνα είμαι Ορθόδοξο Χριστιανό, γνωρίζω πολύ καλά ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία όχι μόνο δεν κάνει προπαγάνδα, ούτε καν πολλέ φορέ υπερασπίζει τον εαυτό τη. Εφαρμόζει την ρίση του Ευαγγελίου όταν δεχτεί ένα χτύπημα στο ένα μάγουλο, γύρισε και το άλλο μέρο του προσώπου σου. Άρα λοιπόν μου κάνει εντύπωση γιατί χρησιμοποιείται αυτή η περίπτωση της ε, Ορθοδόξης Εκκλησίας. Άλλο ένα ερωτηματικό που έχω είναι ότι η Ρωσία αμφισβητεί τις δυτικές αξίες. Ποιες αξίες αμφισβητεί η Ρωσία. Θα ήθελα παρακαλώ και σε αυτό μια απάντηση. Και τέλος αναφέρεται ότι η Ρωσία παραποιεί την ιστορία. Ποια ιστορία παραποιεί. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Επιτελείο. Δεν νομίζω ότι είμαστε τόσο επιθετικοί, ούτε έχουμε επιλέξει να είμαστε αντίπαλοι και όχι εταίροι με κάποια άλλη χώρα. Η κυρία τώρα μπορεί να σας πει ίσως κάτι περισσότερο. Ήταν η συγγήτριά μας το παρελθόν για την ε, συνολική παγκόσμια στρατηγική μας και αυτό είναι ένα θέμα που μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ακριβώς αυτό ήταν που ήθελα να πω, ότι θεωρώ ότι η έκθεση της κυρίας Φωτίγκα είναι τμήμα της συμβολής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην προετοιμαζόμενη έκθεση από την κυρία Μογκερίνη για την παγκόσμια στατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα θέματα ασφάλειας και εξωτερικής πολιτικής. Ζούμε σε ένα ψηφιακό κόσμο. Είμαστε διασυνδεδεμένοι και αλληλοεξαρτημένοι. Το θέμα που μας απασχολεί σήμερα είναι πώς θα βρούμε την δύσκολη αυτή ισορροπία μεταξύ ελευθεριών των μέσων ενημέρωσης και του ελεύθερου ανταγωνισμού. Γιατί αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να μιλήσουμε για ελευθερία ανταγωνισμού αν δούμε εταιρείε όπως η Russia Today ή το Sputnik που έχουν κρατική χρηματοδότηση η οποία είναι σημαντική. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντική η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όχι μονάχα να κάνει μια έρευνα για αυτές τις μορφές υβριδικού πολέμου και πολέμου πληροφόρησης, αλλά η έρευνα αυτή Θα πρέπει με τον τρόπο αυτό να δούμε επίσης και με την έρευνα αυτά πώς μπορούμε να προωθήσουμε τις ευρωπαϊκές ιδέες και να τις χρηματοδοτήσουμε γιατί χωρίς τη χρηματοδότηση δεν θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τις ε, αντίπαλες ιδεολογίες. Και κάτι άλλο το οποίο για μένα είναι πολύ σημαντικό είναι το εξή. Πρέπει να αποδώσουμε μεγαλύτερη προσοχή στην παιδεία. Πώς να αναλύουμε την πληροφορία και πρέπει να είναι μια διαδικασία εκπαίδευσης διαβίου. Δεύτερον, πρέπει να σκεφτούμε πώς θα ενισχύσουμε τα ευρωπαϊκά δίκτυα πληροφορίας και πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την γνώση που έχουμε ήδη συσσωρεύσει σε άλλους διεθνείς οργανισμούς και ιδίως εδώ θέλω να αναφερθώ στο εξαιρετικό αυτό κέντρο του ΝΑΤΟ στην Ρήγα. Υπάρχουν όμως και άλλοι φορείς που μπορούν να παίξουν αυτό τον ρόλο. Τέλος έχουμε στο θέμα της ε, παράνομης χρηματοδότησης που περνούν μέσα από διάφορους διάβλους και χρησιμοποιούνται για να τροφοδοτούν αυτούς τους υβριδικούς πολέμους πληροφορίας. Όχι μόνο τα κρατη πρέπει να έχουν υπηρεσίες συλλογής πληροφοριών που εξετάζουν τα θέματα αυτά και ξέρουμε ότι τα κράτη-μέλη το κάνουν αυτό, αλλά πιστεύω ότι θα πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μας στη δημιουργία μιας ε, υπηρεσίας πληροφοριών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα μπορεί να ανοιχνεύει τις παράνομες χρηματοδοτήσεις που πηγαίνουν σε δημοσιογράφους και μίχιο που προσπαθούν να παραμορφώσουν και να στρεβλώσουν την ε, επακριβή και τίμια επικοινωνία. Είναι πολύ εύκολο λοιπόν το να κάνει κανείς πλήση εγκεφάλου στον κόσμο. Και είναι απαραίτητο να κάνουμε ό,τι χρειάζεται για να προστατεύσουμε τις αξίες μας. Αυτό είναι το μεγαλύτερο καθήκον μας. Ευχαριστώ. Thank you very much. Uh, Σας ευχαριστώ πολύ Σάνδρα και θα ξαναδώσω το λόγο στην συγκεκριά μου στην κυρία Φωτή. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους αυτούς οι οποίοι έλαβαν το λόγο σήμερα και ήταν συνομιλητές μου σε αυτή τη συζήτηση, η οποία είναι μια πάρα πολύ σημαντική, διότι χάρη σε αυτήν μπορούμε να κρίνουμε ποιε είναι οι δυνατότητε ανταλλαγή απόψεων σε σχέση με αυτή την έκθεση, όπως ανέφερα προηγουμένω. Η δομή των θεμάτων αυτών και η σύνθεση όλων των θέσεων δεν ήταν τόσο εύκολη. Υπάρχουν στοιχεία που μπορούν να υποστηρίξουν πολλές απόψεις, αλλά θα πρέπει να έχουμε μια σωστή βάση συζήτησης. Εγώ εκτιμώ ιδιαίτερα την, ε, το σχέδιο γνωμοδότησης της Επιτροπής Προϋπολογισμού, πολιτισμού, που μας παρέχει μια, ένα νέο μια νέα οπτική γωνία για τη, για τη σκέψη μας στην έκθεση αυτή, είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό για να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις ιδέες. Με ενδιαφέρε ιδιαίτερα το σχόλιο αυτό για την αναγκαιότητα να αντιμετωπίσουμε τον υβριδικό πόλεμο και τα υβριδικά εργαλεία και είμαι πάντα έτοιμη να εξετάσω αυτό το θέμα και στο μέλλον σε συναντήσεις με τους σκιώδεις εισηγητές που θα γίνει στην επόμενη σύνοδο του Στρασβούργου και στην οποία προσβλέπω κιόλα. Θέλω ευχαριστήσω τους συναδέλφους που με υποστήριξαν στο θέμα αυτό και βασίζομαι στη βοήθειά σας για να βελτιώσω την έκθεσή μου με τα σχόλιά σας, επιτρέψτε μου και μία ακόμα φορά να αναφέρω το θέμα της στρατηγικής α, πληροφόρησης και επικοινωνίας που προέρχεται από το Κρεμλίνο. Μερικοί θα θέλανε ίσως να χρησιμοποιήσουν να ε, χρησιμοποιήσουν και αυτή το σύστημα του Πούτιν για να μας χειραγωγήσουν στη Δύση. Και πρέπει στην έκθεσή μας να συνδεθεί και με τους κοινούς που προέρχονται από τη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική, κυρίως στη στρατηγική επικοινωνία από τον ΤΑΕΣ. Είτε το θέλουμε, είτε δεν το θέλουμε, υπάρχουν πολλές οντότητες σήμερα οι, οποίοι, οι οποίες στρέφονται εναντίον μας και πρέπει να τα κατανοήσουμε όλα αυτά. Να καταλάβουμε ότι είναι πολύ σχηλής αυτή η απειλή και χρειάζεται να έχουμε διαφορετικά εργαλεία για να αντιμετωπίσουμε αυτές τις απειλές, αλλά δεν θα πρέπει να παραμείνουμε αφελείς και αδρανείς στην αντιμετώπιση αυτών των άλλων απειλών, γιατί απειλές είναι. Και απαντώντας στα σχόλια του κυρίου Φρόιντ για την ενδεχόμενη διαφορά μεταξύ της Πολωνίας και της Πορτογαλίας ως ε, αντικείμενα ρωσικής προπαγάνδας. Μα το λέει η έκθεσή μου ότι οι δράσεις οι οποίες έχουν αναλυθεί από τη ρωσική πλευρά είναι ιδιαίτερα στοχευμένες προς το ακροατήριο συγκεκριμένων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διαφέρουν από χώρα σε χώρα. Και είναι προφανώς μεγαλύτερη προσπάθεια, θα έλεγα, η οποία έχει αναλυθεί έναντι της Πολωνίας. Παρ' όλα αυτά είμαστε εμβολιασμένοι, θα έλεγα, μέσα σε εισαγωγικά, από αιώνες που μας έχουν συνηθίσει στη ρωσική στάση. Δεν είναι τυχαίο λοιπόν ότι μεταξύ των ανθρώπων που έχει βάλει ο Πούτιν στη μαύρη λίστα υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός Πολωνών. Είναι διαφορετική λοιπόν η κατάσταση σε κάθε χώρα ενδεχομένω, αλλά η συνολική διαδικασία είναι ότι οι ρωσικές ενέργειες κατευθύνονται και στην ίδια τάξη μεγέθους προς όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και θυμηθείτε την ιστορία της ε, Λίζας στη Γερμανία, παρουσιάστηκε αυτό το θέμα και πολύ σωστά. Ευχαριστώ κυρία Φωτίγα για το για τα συμπεράσματά σας. Θα υπάρξει συζήτηση και διαπραγμάτευση μεταξύ των ε, σχεδόν συγγητών. Είναι φανερό ότι υπάρχουν διαφορετικές απόψεις και είναι απαραίτητο να συγκεκριμενοποιηθούν οι απόψεις για το πώς μπορούμε να είμαστε λειτουργικοί και πώς εμπλέκονται τα θρησκευτικά θέματα και σε αυτή τη συζήτηση. Καλή τύχη. Σας υπενθυμίζω σε όλους ότι οι προθεσμίες της τροπολογίας για το σχέδιο αυτό είναι στις 26 Μαΐου σε δύο μέρες. Όλοι αυτοί οι οποίοι θα υποβάλουν τροπολογίες παρακαλώ κάντε το το συντερότερο. Και η επόμενη εξέταση αυτής της έκθεσης είναι 27 Ιουνίου στην 12 ε, Ιουλίου στην ΑΦΕΤ και Σεπτέμβριο στην Ολομέλεια. Δύο ανακοινώσεις και μία αλλαγή της ημέρησης διάταξης. Θα συζητήσουμε τώρα για την επίσκεψη της Επιτροπής μας στη Βοσνία Ζεγοβίνη ε, την προηγούμενη εβδομάδα, γιατί ήταν ένα θέμα που το αναβάλαμε από την πρωινή συνεδρίαση. Και δεύτερον, απόψε, ορισμένα από εσά έχετε προσκληθεί ως αντιπροσωπεία, η αντιπροσωπεία για την ε, Ουκρανία θα δει ένα έργο, υπάρχει μια πρόσκληση για το έργο ο χειμώνα καίγεται, που είναι η παρουσίαση των γεγονότων του Μαϊντάν, θα ξεκινήσει κάποτε, κάπως νωρίτερα στις 7.30 ε, ξεκινά στο Μποζάρ και είσαστε όλοι προσκεκλημένοι. Αν θέλετε, πέστε μας αν θέλετε να πάτε. Και τώρα έρχομαι στο σημείο αυτό για την επίσκεψη στη Βοσνία Εζεγοβίνη. Πήγαμε στο Μόσταρ και στο Σεράγεβο την Τετάρτη και την Πέμπτη. Ήταν η πρώτη επίσκεψη της Άφρετ στη Βοσνία Εζεγοβίνη μετά από την ε, υποβολή μιας επίσημης αίτησης για προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση 15 Φεβρουαρίου του 2016. Θυμόσαστε πόσο σημαντικό ρόλο έχει παίξει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τη δημιουργία ενός θετικού κλίματος για την θετική υποδοχή αυτής της αίτησης, ιδίως σε επίπεδο Συμβουλίου και την υποστήριξη που πήραμε και από την Κομισιόν και την κυρία Μογκερίνη καθώς και τον Επίτροπο κύριο Είχαμε λοιπόν αυτές τις ε, συζητήσεις στο Μοστάρ, μια από τις μεγαλύτερες πόλεις μετά το Σεράγεγο στη Βοσνία Ζεγοβίνη, με κυριότερο θέμα την εφαρμογή του συνταγματικού δικαστηρίου από το 2010 για να μπορέσει να προετοιμάσει το, πλαίσιο, το νομικό πλαίσιο για τις τοπικές εκλογές. Δυστυχώς δεν είχαν γίνει τοπικές εκλογές μέχρι το 2008 με τις, και δεν έγινε τελικά με τις τοπικές αυτές εκλογές που θα γίνουν στις αρχές Οκτώβριου, προϋποθέτει αυτό μια συμφωνία των πολιτικών κομμάτων. Στο Εγώ συναντηθήκαμε με τον πρόεδρο της Προεδρίας, τον κύριο Ζεμπέκοβιτς, τον πρόεδρο Σβίζης του Συμβουλίου των Υπουργών που είχε έρθει στην Επιτροπή μας στο Στρασβούργο πρόσφατα και επίσης τους ε, πρωθυπουργούς της Ομοσπονδίας και της Ρεπούμπλικας Σέρψκα. Συναντήσαμε επίση του ομολόγους μας από το Κοινοβούλιο της Βοσνία Ερζεγοβίνη, τους συναδέλφου μας από την ε, Αντιπροσωπεία σταθεροποίηση και ε, Σύνδεσης, μέσω στόχο να στείλουμε και πάλι το μήνυμα ότι πρέπει να εγκριθούν οι κανόνες ε, διαδικασίας αυτής της Επιτροπής στην επόμενη συνεδρίασή μας του Ιουνίου στο Στρασβούργο. Είχαμε επίσης εκτενείς επαφές με τους ε, Ευρωπαίους διπλωμάτες, με τον κύριο Βίγκεμαρ που είναι ο ειδικό εκπρόσωπος τη Ευρωπαϊκής Ένωσης, με ΜΚΟ και τα λοιπά. Φυσικά έχει η χώρα αυτή όχι μονάχα την προτεραιότητα της εφαρμογή του θεματολογίου μεταρρύθμισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και την ανάγκη να δημιουργήσει ένα μηχανισμό συντονισμού και την ε, τροποποίηση συμφωνίας για να σύνδεση για να λάβει υπόψη την ε, είσοδο της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε θετικά αποτελέσματα από το, την απογραφή που οργανωθεί το 2013 και είναι απαραίτητη για να έχουμε σωστέ τοπικέ εκλογέ τον Οκτώβριο. Το μήνυμα μα δεν είναι μόνο να ενθαρρύνει τι αρχέ να προωθήσουν τι ευρωπαϊκέ μεταρρυθμίσει, αλλά να εξασφαλίσουν και τη συνεκτικότητα τη χώρα, γιατί υπάρχουν ορισμένε αποσχιστικέ τάσει οι οποίε αναδύονται κάθε τόσο στο τμήμα τη χώρα που ονομάζεται Ρεπούμπλικα Σέρψκα όπου ο κ. έχει προτείνει ήδη δύο δημοψήφισματα, τα οποία δεν έχουν γίνει, αλλά είδαμε πώς με, κάποιο, με έναν τρόπο που είναι απαράδεκτο. έχει εμποδίσει ενέργειες ατόμων που είχαν επισκεφτεί το Ευρωπαϊκό μας Κοινοβούλιο, κάτι άλλο το οποίο είναι απαραίτητο είναι να εξασφαλίσουμε ότι θα εξεταστεί από το Συμβούλιο για τις υποσχόλησεις της Βοσνία Ζεγοσκοπίνης. Ελπίσουμε ότι θα μπορούσε να δοθεί το καθεστώ τη χώρα υποψηφίου μέσα στο 2017 και ελπίζουμε ότι θα μπορέσουν να ληφθούν κάποιε τέτοιε θετικέ αποφάσει κατά τη διάρκεια τη Σλοβακική προεδρία Και τώρα θα δώσω το λόγο στον Κρίστιαν Πρέντα, τον εισηγητή μα, ο οποίο έχει συντάξει μια εξαίρετη έκθεση που εγκρίθηκε πριν από δύο μήνε και μπορεί να μα πει και περισσότερα για τη διαδικασία μεταρρυθμίσεων μετά από την επίσκεψή μας στο Μόστρα και το Σεράγεβο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, ο κ. Σουάπλενκο έκανε μια πολύ ολοκληρωμένη παρουσίαση των όσων πράξαμε εμείς στην Φωσνία εντός μιας εβδομάδας. Ουσιαστικά ξεκινήσαμε από το Μουστάρ. Αρχικά όταν σχεδιάζαμε το πρόγραμμα της επίσκεψης, σκοπός ήταν να πάμε στο Μοστάρ ε, για να συγχάρουμε επιτέλους τις πολιτικές δυνάμεις της Βοσνίας Ερζεγοβίνης ε, για τη σύναψη μιας συμφωνίας ε, που θα μπορούσε να οδηγήσει σε τοπικές εκλογές και στο Μοστάρ. Δυστυχώς οι διαπραγματεύσεις που φαίνονταν θετικές δεν περατώθηκαν με καλό αποτέλεσμα. Έτσι λοιπόν εμείς εκεί Ακούσαμε τους ε, κύριους πολιτικούς ε, ηθήνοντες, ε, το SDA, STZ, το SDP, το DF. Συζήτησαμε με αυτές τις σημαντικές πολιτικές δυνάμεις της χώρας και προσπαθήσαμε να καταλάβουμε γιατί οι πολιτικές εκλογές, οι τοπικές, που έπρεπε να λάβουν χώρα παντού στη Βοσνία Ζεγοβίνη, αλλά όχι στο Μοστάρ, να θυμίσω ότι είχε γίνει και παλιότερα αυτό και αυτό που μας εξέπλεξε είναι ότι μας είπαν είναι ευθύνη της διεθνούς κοινότητας να βρει μια λύση. Εμείς ε, ανταπαντήσαμε λέγοντας ότι η Βοσνία πρέπει, η Βοσνία πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες της σε πολιτικό επίπεδο στον αφορά το Μοστάρ. Δώσαμε δηλαδή ένα χειρό μήνυμα στους πολιτικούς συνθήνοντες ε, και στην συνάντηση που είχαμε τον πρόεδρο Ζαρμπαϊκοβίτς ε, για το πόσο σημαντικό είναι να γίνουν εκλογές στο Μοστάρ. Δεύτερον, συζητήσαμε εκτενώς ε, στη διάρκεια των διαφορών συναντήσεων μας στο Σεράγεβο για το ζήτημα που αποτελεί και σημαντική προσδοκία των αρχών στην απάντηση για τη... Απάντηση δηλαδή για την υποβολή, στην υποβολή υποψηφιότητα. Ε, είπαμε λοιπόν ότι είναι αναγκαίο να εκπληρωθούν οι τρει δεσμεύσει ε, που είναι πολύ σαφεί. Ο Αντρέ ανέφερε ήδη. Ο μηχανισμό συντονισμού που έχει καθυστερήσει. Η προσαρμογή της Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης ε, και σε σχέση με την Κροατία και φυσικά και ε, το άλλο θεματολόγιο, σημεία πολύ σημαντικά. Αυτό το μήνυμα λοιπόν έδωσε η αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο κ. Βέγερμακ, ε, κυρίως, ε, και θα παραλάβουμε πολλάκες. Και είχαμε και την σοβαρή βοήθεια της πολωνικής αντιπροσωπείας στην επίσκεψη αυτή. Τώρα, όσον αφορά τις επαφές ε, με τους πολιτικούς ηθήνοντες, πρέπει να αναφέρω το γεγονός ότι είχαμε την ευκαιρία να συναντηθούμε με τους δύο ε, πρωθυπουργούς Ναβαλίτς Τζιάνοβιτς και στη διάρκεια αυτή της συνάντησης εγώ παρουσίασα στην κυρία Τζιάνοβιτς ε, ένα κομμάτι της έκθεσης που υιοθετήθηκε θα θυμάστε μεγάλη πλειοψηφία από το κοινοβουλίο μας και που αφορούσε την Ρεπουμπλικά Σέρψκα. Η αντίδρασή της ε, δεν ήταν ιδιαίτερα φιλική πρέπει να πω. Χαρακτήρισε επιφανειακή την έκθεση αυτή και και μεροληπτική ε, και δεν έδειξε ιδιαίτερη διάθεση να συνεργαστεί μαζί μας. Και εμεί είπαμε λοιπόν, ότι θέλουμε η Ρεπούμπλικα Σερψικά και οι αρχές της ε, να συμμετέχουν και αυτές σε αυτή την προσπάθεια, την κοινή προσπάθεια όλων των ε, ηθινόντων ε, στην πορεία αυτή της Βοσνία Ερζεγοβίνη προ την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εγώ λοιπόν επαναλαμβάνω αυτή την έκκληση για συνεργασία στου ηθινοντέ τη Ρεπούμπλικα Σερψικά. Είχαμε κάποιες, κάποια καλά νέα όσον αφορά την απογραφή αλλά και το πώς θα χρησιμοποιηθεί, δηλαδή τι μεθοδολογία θα χρησιμοποιηθεί για τα αποτελέσματα, για τον υπολογισμό και την δημοσίευση των αποτελεσμάτων. Έκτοτε, δυστυχώ, είχαμε κάποιες εξελίξεις ε, αποθαρρυντικέ. και πάλι εκ μέρους της Ρεπομπλικά Σέρψκα. Κάτι σημαντικό που αναφέραμε και το οποίο είναι σημαντικό για τη χώρα αυτή είναι το ζήτημα της καταπολέμησης διαφθοράς και του γεγονότος ότι πέραν των προσπαθειών των ε, θεσμών που είναι σημαντικές. Ε, κάποιοι εισαγγελεί δεν φοβούνται να διεκπαιρεώσουν ε, φακέλους που σχετίζονται με πολιτικούς ευθύνοντες. Ε, πρέπει και τα ίδια τα πολιτικά κόμματα να αναλάβουν την ευθύνη αυτή του αγώνα κατά της ε, διαφθοράς. Τέλος, ε, δώσαμε το μήνυμα ότι υπάρχει μια ανάγκη να δούμε και τις απόψεις των συναδέλφων βουλευτών της Βοσνίας όσον αφορά τις εργασίες για το SPSC. Σε ορισμένες μέρες πρόκειται να γίνει μια συζήτηση και ο πρόεδρος μας, ο κ. Σέλμαρ Μπρόκ, ο οποίος μόλις ξαναήρθε στην έτσι, με τον συνάδελφο Πίτσουλα. Κύριε Πρόεδρε, για σας μιλάω. Ο πρόεδρος μας λοιπόν, ο κ. Μπρόκ και ο κ. Τονίνο Πίτσολα μια επιστολή εκ μέρου τη Επιτροπής μας όσον αφορά την υιοθέτηση αυτών των κανόνων. Έλεγα λοιπόν ότι εμείς υπενθυμίσαμε στους συναδέλφους μας βουλευτές εκεί ότι είναι σημαντικό να υιοθετήσουν μια λογική θέση ώστε ε, το όργανο αυτό που διευκολύνει τη συνεργασία μεταξύ Βόσμων Βουλευτών και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να υιοθετήσει στην επόμενη ε, συνεδρίαση που έχει προγραμματιστεί τον Ιούνιο, αρχές Ιουνίου. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Πιστεύω λοιπόν ότι ήταν πολύ επικοδομητική η επίσκεψη και ευχαριστώ και την ε, αντιπροσωπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης επί που μας βοήθησε ιδιαίτερα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ε, παρουσίαση των νέων από την επίσκεψη στην Βοσνία. Να ακούσουμε και μια φωνή από την Κροατία, την κυρία Σβίτσια. Σα ευχαριστώ. Συμμετείχα μόνο την πρώτη ημέρα στην επίσκεψη στο Μοστάρ. Δεν έχω να πω και πάρα πολλά λοιπόν. Σύμφωνα με την άποψή μου, υπάρχει μια διαφορά όταν μιλάμε εδώ στο Κοινοβούλιο, όταν κάνουμε διακηρύξεις και δηλώσεις και υπάρχει διαφορά όταν βλέπουμε την κατάσταση επιτόπου. Είναι πολύ διαφορετικό. Και αυτό που με εντυπωσιάζει όλος ιδιαίτερος είναι ότι πολιτικός μιλώ για τους τοπικούς πολιτικούς του Ομοστάρ, δεν μπορούν να συμφωνήσουν ε, για τις εκλογές. Αν δεν μπορεί να υπάρξει λοιπόν πλειοψηφία στην κοινοβουλευτική συνέλευση στο Σαράγεβο σε ό,τι αφορά το σταγματικό δικαστήριο, και χρειάζεται μάλλον να αποφανθεί το συνταγματικό δικαστήριο. Το θέμα είναι πώ θα προχωρήσουν σε πιο σοβαρά ζητήματα. Αυτό αναρωτιέμαι. Αν και πάντα είμαι υπέρ τη Βοσνία Ερζεγοβίνη, πάντα ήμουν, είμαι πάντα της, υπέρ τη ένταξή του στο ευρωπαϊκό έργο. Τέτοια ζητήματα όμω πραγματικά με προβληματίζουν. Θα πρέπει να αλλάξουν λοιπόν το εκλογικό δίκαιο. Δεν μπορούν να αλλάξουν το εκλογικό δίκαιο χωρίς να εφαρμόσουν τις αποφάσεις αυτές του συνταγματικού δικαστηρίου. Ας δούμε λοιπόν τι θα γίνει. Από ό,τι άκουσα η επίσκεψή σας στο Σαράγεβο ήταν καλή και προσβλέπουμε σε μια πιο προοδευτική προσέγγιση. Σας ευχαριστώ πολύ και ας συνεργαστούμε λοιπόν για τη Βοσνία Ζεγοβίνη. Ο επόμενο, ο πρόεδρος. Μία σύντομη παρατηρήση θα ήθελα να κάνω. Και αυτό κατέστη σαφέ σε ό,τι αφορά την επίσκεψη στο Μόστα, παρά το γεγονό ότι εγώ προσωπικά δεν μετέβησα εκεί παρά μόνο στο Σαράγεβο. Στη Βοσνία Ερσεγοβίνη είναι ιδιαίτερα σημαντικό το θέμα αυτό, όχι όμως μόνο στη Βοσνία Ερσεγοβίνη. Στις χώρες αυτές λόγω φόβου για το παρελθόν δεν έχουν ε, συχνά οι άνθρωποι την τόλμη να ταινίσουν το μέλλον και μπλοκάρουν ε, αλλήλους προκειμένου να εμείνουν στις σημερινές τους θέσεις. Και έτσι λοιπόν ε, α, αναδύεται πάντα το παρελθόν και η Βοσνία Ζεγοβίνη και η κατάσταση που επικρατεί εκεί αποτελεί ένα μικρό κλίμα, ένα μικρό κόσμο του φαινομένου αυτού. Και στο, το αποτέλεσμα είναι ότι επιδεινώνονται οι συνθήκες διαβίωσης του κόσμου εκεί. Δεν βελτιώνονται. Όσο λοιπόν δεν υπάρχει αυτή η έννοια της εμπιστοσύνης, ε, της αισιοδοξία για το μέλλον, θα μείνουν κολλημένοι σε αυτή τη φάση. Και γι' αυτό είναι υπεύθυνε και οι τρεις ε, κοινότητες, σε διαφορετικό βαθμό ενδεχομένω. Θα πρέπει να βρούμε λοιπόν ένα νέο τρόπο προσέγγισης ως προς το περιεχόμενο, ως προς την αντιμετώπιση. Και ήταν ε, ενδιαφέρουσα συναντήσεις με τον ε, Πρωθυπουργό της Ομοσπονδίας και της Ρεπούμπλικα Ρεπούμπλικα Πρόκειται για μια νέα γενιά. Ε, επί του περιεχομένου δεν έχει αλλάξει κάτι, αλλά είχα την εντύπωση ότι η σχέση μεταξύ των ατόμων ήταν πιο επικοδομητική πλέον από ό,τι στο παρελθόν. Η στάση μεταξύ τους. Ελπίζω να μην ε, αυταπατώμε. Και θεωρώ ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό μήνυμα στη τελική ανάλυση. Ξέρουμε ότι η χώρα θα μείνει ενωμένη και ότι θα υπάρχει αυτή η προοπτική ευρωπαϊκή. Ελπίζω να μην είναι κάτι το ψευδές ε, η ευρωπαϊκή αυτή προοπτική προκειμένου να διατηρηθεί το status quo αλλά να, αποτελεί μια πραγματική δυνατότητα. Δεν είμαι βέβαιος να σας πω. Είναι κάτι τεχνητό για να τηρηθεί το ευρωπαϊκό πλαίσιο γιατί δάλλως ε, θα σπάσουν προς όλες τις κατευθύνσεις οι δυνάμεις αυτές. Και νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να το δείξουμε και να το πραγματευτούμε ανοιχτά μαζί τους και να μην το κρύβουμε πίσω από διπλωματικές κουρτίνες το οποίο θεωρώ ότι το κάναμε υπερβολικά μακρύ χρονικό διάστημα. Θα πρέπει λοιπόν να δημιουργηθεί και η νοοτροπία, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τη νέα γενιά ότι τους κατανοούμε. Ιδάλλως τα πράγματα θα κινηθούν προς τη λάθος κατεύθυνση. Δεν μπορεί να παραμείνει αυτή η κατάσταση. Δεν ε, μπορεί να παραμείνει έτσι η κατάσταση, γιατί σε 20 χρόνια θα βρισκόμαστε ακριβώ στο ίδιο σημείο σε ό,τι αφορά την ευρωπαϊκή προοπτική. Και αυτό φυσικά δεν έχει και δεν εξυπηρετεί κανένα συμφέρον, ούτε τα δικά μα ούτε τα συμφέροντα τη περιοχή. Γι' αυτό ρωτιέμαι πως η επόμενη κοινή συνάντηση με του. Ε, πρωθυπουργούς ε, του, της Ομοσπονδίας και της Ρεπουμπλικής Έλψικα μπορεί να λάβει χώρα στην Πάνια Λουκά. Αυτή είναι η διαφορά. Γιατί πολλά πράγματα τέτοια θα έπρεπε να τα κάνουμε. Γιατί και οι δύο δήλωσαν ότι ήταν δεθμένοι να το κάνουν αυτό. Πολύ απλά για να αλλάξουν και λίγο οι νοοτροπίες και οι αντίληψεις. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να κάτσουμε να το σκεφτούμε. Να ευχαριστήσω τους συναδέλφους που συμμετείχαν και θα ήθελα στο σημείο αυτό να κλείσω τη συνεδρίαση και να, περνάμε, να περάσουμε στη συνεδρίαση του Προεδρείου. Στις 2 Ιουλίου είναι η επόμενη συνάντηση. Την 2 Ιουνίου είναι η επόμενη συνεδρίαση. Την άλλη Πέμπτη. Και παριλαμβάνει η ημερήσια διάταξη. είναι η μέρα που δεν θα έρθει καθόλου το ΕΛΚ. Έχει εξωτερική συνάντηση. Αν δεν είναι απόλυτα απαραίτητο να γίνει συνεδρίαση στις 2 Ιουνίου, θα πρότεινα να την διαγράψουμε και να το ξαναπούμε στις 13-14 Ιουνίου κατευθείαν. Και στις 6 Ιουνίου έχουμε βεβαίως, βεβαίως μία συνάντηση στο Στρασβούργο. και μήπω εκεί μπορούμε να κοιτάξουμε κάποια απαραίτητα ζητήματα τα οποία θα κοιτάξουμε στις δύο του μηνό. Συμφωνείτε. Γιατί παραδοσιακό πώ ε, δεν είναι πολύ συμμετέχοντε σε αυτέ τι συναντήσει τη ε, μισή ημέρα, τη Πέμπτη. Ε, ξέρετε γιατί, γιατί όλοι πηγαίνουν στι εκλογικέ του περιφέρειες και ο κύριο Τάνοκ θα έχει και χρόνο να σκεφτεί. Σας ευχαριστώ πολύ και τη στις σα.